Καλημέρα σας αγαπητοί συναδελφοί, σας καλωσορίζω θερμά. Να σας παρουσιάσω και ένα ε, καινούριο, μάλλον δύο καινούριου βοηθούς, την Καταρίνα Χέσλεβικ και τη Σαντρίν Κουτιέ που είναι τα νέα μέλη της γραμματείας και εμπλουτίζουν τη γραμματεία της Επιτροπής του Προπολογισμού. Άρα είμαστε αρκετοί τώρα. Δεύτερο, έχετε σε ό,τι αφορά οι προβλήματα με τη Μέσια διάταξη. Παρακαλώ, κύριε Φρόιντ. Όχι σε ό,τι αφορά τη Μέσια διάταξη. Απλά σύντομα θα ήθελα να συγχαρώ για την πολύ επιτυχημένη επιστολή που γράψατε εξ ονόματος όλων μας και αποφεύθηκε η ε, σπατάλη πάρα πολλών ε, χρημάτων ε, των φορολογουμένων για, τις, για τους επιτρόπους. Όχι, δεν το έκανα για κάποιο συγκεκριμένο, το έκανα για όλους, λέει η Πρόεδρος. Όταν πήρα αυτή την είδηση ε, και πριν μπορέσω να με κανέναν ε, και ζήτησα, τη, ζήτησα συγγνώμη γιατί δεν μπορούσα να ενημερώσω, έγραψα αυτή την επιστολή. Συνήθως το κάνω αφού έχω ε, συζητήσει με τους συντονιστές. Δεν υπήρχε όμως δυνατότητα να μιλήσω με κανέναν και γι' αυτό δεν ακολουθώ αυτή τη συνήθεια διαδικασία. Πάντως, για αύριο έχω να σας πω ότι ε, έγινε μια μεγάλη, είχαμε μια μεγάλη επιτυχία σε ό,τι αφορά την εισαγγελία ε, και είχαμε διαπραγματευτεί με τη Λίμπε και την Κοντ ε, και η κυρία είναι η πρώτη Ρουμάνα που πλέον αναλαμβάνει μια κορυφαία θέση στο, στο, ως επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι μια πολύ ικανή γυναίκα και νομίζω ότι ε, είναι το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Έχει στελεχωθεί με τον καλύτερο τρόπο ε, το γραφείο της, Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Θέλουμε να μπορούμε να διερευνούμε τα θέματα του διεθνούς εγκλήματος, της, ε, του ξεπλήματος κλίματος κτλ. Ήταν λοιπόν μια μεγάλη επιτυχία αυτό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας πω κάτι που ξέρετε πολύ καλά, να χαμογελάτε και να είστε έτσι ευπροσίγουροι, διότι μας ε, παίρνουν οι κάμερες. Επίσης για τη διερμηνία έχετε τις γλώσσες, βλέπετε τις καμπίνες, έχουμε αρκετέ γλώσσες και περνάω τώρα στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης που είναι η απαλλαγή για το 2017 δεύτερη έκθεση για τον Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αποστήριξη Ασύλου ΕΑΣΟ. Καταρχάς να δώσω το λόγο στον εισηγητή. thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το έχουμε πει αυτά τόσες φορές ε, με ευκαιρία διάφορες συναντήσεις, οπότε δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Αφού τα έχουμε πει, ας πάμε στην ψηφορία. Ωραία. Έχετε όλοι τις κάρτες ψηφοφορίας. Good. Wer also für Petri Όποιος θέλει λοιπόν να στηρίξει την πρόταση ε, Πέτρη Σαβάρμα, βέβαια υπάρχουν ε, κάποιες διακοιμάσεις, όποιος δεν θέλει, δηλαδή ε, ψηφίζει υπέρ του Σαβάρμα και όποιος θέλει την, να δοθεί απαλλαγή ψηφίζει κατά. Es geht jetzt zu Antrag 1, Petri äh, Savarma. Δηλαδή, όποιο θέλει να δώσει απαλλαγή θα ψηφίσει κατά τη πρόταση Σαβάρμα. Έχει τι κάρτε σα ή να ψηφίσουμε διανατάσεω. Ποιο είναι κατά. αποχές Άρα δεν δίνουμε απαλλαγή, δεν χορηγείται απαλλαγή. Ψηφίσατε υπέρ την πρόταση Σαββάτ. Okay, we have to do a... Ε, από ό,τι μου λένε εδώ, πρέπει να ψηφίσουμε μονομαστική κλίση για την απαλλαγή. Mm. Συγγνώμη, είναι η πρώτη φορά που το κάνω, δεν είμαι και τέλεια, με συγχωρείτε. Ποιο είναι υπέρ, λέει η πρόεδρο. Α, όχι, με συγχωρείτε, λέει η πρόεδρο. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, με συγχωρείτε, λέει η πρόεδρο. Okay. 21. 21 ψήφοι υπέρ, καμία κατά 6 αποχές. Περνάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος. Στην πρώτη παράγραφο. Τροπολογία 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Τροπολογία 3. Ψήφι πέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4. Μάλλον παράγραφος 5. Τροπολογία 4. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. Παράγραφος 6. Τροπολογία 5. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7. Τροπολογία 6. Ψήφι πέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Compatible συμβατή υπέρ της 7. Κατά. Να ελέγξουμε. Εντάξει, ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 16 προς 10. 16 προς 10. 8. Μαρία Γαμπρίν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Παράγραφος 8, τροπολογία 9. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Συγγνώμη, 9. Τροπολογία 10. Ψήφι ΠΕΡ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Τροπολογία 11. Ψήφι ΠΕΡ κατά αποχές απορρίβεται τροπολογία 12 12 ναι γιατί δεν, ήταν, δεν, δεν προηγουμένη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 13 στη 10 πάντα ψηφιπέρ κατά να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 7 ψηφίπερ υπέρ, 16 κατά και 3 αποχές. Τώρα, παράγραφος 10α, ε, τροπολογία 14, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 10β, τροπολογία 15, ψήφι υπέρ. Α, με συγχωρείτε, λέει πρόεδρος, έχει εγκριθεί προηγούμενη, δεν το είχα δει, άρα αυτή δεν την ψηφίζουμε. Πάμε στο 10C, τροπολογία 16, ψήφι υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε, πιστεύετε, εντάξει, ας ελέγξουμε. Αν και νομίζω ότι όλοι πέρυνε. Πέρας ψηφοφορίας. Ναι, 26 ψήφοι πέρα όλοι. Τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 25 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. Και καμία ψήφος κατά. Η πρεμιέρα μου ήταν, τώρα θα βελτιωθώ σιγά σιγά. Το παρθενή, η παρθενική μου ψηφοφορία. Πάμε στο επόμενο σήμα της μερίσιας διάταξη που είναι απαλλαγή. Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεύτερο σχέδιο έκθεση, Ζαμπέλ Γκαρθία Μουνιώθ. Η συγκίτρια δεν ξαναθέλει το λόγο. Ακούστε, όπως και ο κ. Σαρβαμά ε, θα πω και εγώ ότι τα έχω πει ε, στην προηγούμενη συνέδρια Επιτροπής ε, ό,τι είχα να πω, άρα ας περάσουμε στην ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με την ψηφοφορία. Αν θέλετε να υπερψηφίσετε, κατ' ουσίαν δεν δίδεται απαλλαγή. Αν ψηφίσετε μήνους κατά, δίνεται απαλλαγή. Ψηφίζουμε λοιπόν. Έκλεισε η ψηφοφορία. Θέλετε να πείτε κάτι. «25 υπέρ, κανείς κατά, καμία εποχή. Πάμε τώρα στην πρόταση ψηφίσματος, εδάφιο Α, τροπολογία 1, υπέρ παρακαλώ, κατά, εγκρίνεται. Εδάφιο Β. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Εδάφιο C, τροπολογία 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 1 ή 4 γραπίνη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 παράγραφος 2 υπέρ κατά απορρίπτεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 6, Μαρία Γκραπίνη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 8, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 7, τροπολογία 10, υπέρ, split vote, ε, σε χωριστή ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11, συμβατή, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην προφορική τροπολογία υπαριθμών 1, Μουνιώσα Στέλ, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Η 13 υπέρ παρακαλώ. Κατά Τότε ονομαστική ψηφοφορία πρέπει να ελέγξουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Rejected. Rejected. 12-12. Απορρίφθηκε 12 με 12 είναι το αποτέλεσμα, ισοψηφία. Η 14 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 16 για την παράγραφο 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 17 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν κατάλαβα καλά. Οι σοσιαλδημοκράτες ήταν υπέρ. Υπέρ ήταν. Εντάξει, τότε είναι σαφές, εγκρίνεται. Πάμε στην προφορική τροπολογία. οι δύο μουνιώσα στέλ να ε, βγει η λέξη Europeans από την τροπολογία 17. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 13, τροπολογία 18, Ντανιέλ Φρόντ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 14, τροπολογία 19, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. για την τροπολογία 20 ε, τροπολογία ή ε, ζητάτε προφορική ψηφοφορία και γι' αυτό ψηφίζουμε ονομαστικά για την τροπολογία υπερθυμών 20. έκλειση ψηφοφορία. 19 υπέρ, 7 κατά. Προφορική τροπολογία υπαριθμό 3 για την παράγραφο 14α Λούκα Φλένιγκεν. Θα διαβάσω, αναγνωρίζει ότι τα κρατημέλη πρέπει να χρηματοδοτούν τις προεδρίες τους ε, και λυπάται που τον ε, το να καλύπτονται κάποιες δαπάνες ε, από εμάς. Αυτό έχει γίνει πρακτική τα τελευταία χρόνια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε γιατί δεν ξέρω τι έκαναν οι σοσιαλδημοκράτες. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν ε, ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος. Μισό λεπτό. 19 υπέρ, 7 κατά, μία αποχή είναι το αποτέλεσμα της προηγούμενης ψηφοφορίας. Ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Μισό λεπτό. Ναι, με ονομαστική ψηφοφορία. Υπέρ παρακαλώ. Συγγνώμη, τα μπέρδεψα λίγο. Τι, τι ρωτάω ποιο είναι υπέρ. Ε, συγγνώμη, πρέπει να πω ανοίγει η ψηφοφορία και κλείνει. Τι. 26 υπέρ, ένας, ε, μία αποχή, κανένας κατά. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε στο σημείο υπαριθμών 5 της ημερήσιας διάταξης που πρόκειται για τον Γενικό Προεπλογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, χρονιά 2020 για όλα τα τμήματα. Η κυρία Κορίνα Κρετού είναι η συγγήτρια και της δίνω παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η έκθεση είναι περίπλοκη. αφορά τον προϋπολογισμό του 2020 που όπως γνωρίζετε είναι η τελευταία χρονιά του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου και πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πάσχεσαν για αυτή την έκθεση και τους συναδελφούς της Επιτροπής και των πολιτικών ομάδων προσπαθούμε να αντιλήσουμε συμπράσματα από σε στο παρελθόν προσπαθήσαμε να συντάξουμε μια έκθεση που θα είναι στο πνεύμα της συνέχειας και έτσι να γίνει η μετάβαση στο καινούριο πλαίσιο. Τα συζητήσαμε, δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να επαναλάβουμε τη συζήτηση, αλλά να ξαναευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για αυτές τις 22 ε, τροπολογίες. Ας πάμε στην ψηφοφορία. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ τους εισηγητές ε, για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει και θα ήθελα να έρθουμε στην παράγραφο 10α, η τροπολογία 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οι δύο για την 10α πάντα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 3 ε, για το 4α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για το 5 τροπολογία 4 υπέρ κατά εσείς οι σοσιαλδημοκρατές τι είστε υπέρ ή κατά υπέρ είστε. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 7. Για το 5α. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11α. Τροπολογία 8 προφορική τροπολογία αναφέρεται ότι υπάρχει το ανθρωπιστικό στοιχείο σε κάθε θέμα μετανάστευσης ε, που αναγκαστικά θα οδηγήσει σε έκτακτα μέτρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Επαλήθευση. Ναι. Ψηφίζουμε. Mm. Έκλεισε ψηφοφορία. 14 υπέρ, 10 κατά, 3 ε, αποχές και έχουμε μετά την... Ε, όχι, όχι, μισό λεπτό, όχι ακόμα, λέει η πρόεδρος, όχι ακόμα. Η 9 για την 11α υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 για τη 12 υπέρ κατά αποχές πρέπει να παληθεύσουμε Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. 20 υπέρ, 6 κατά. Ε, τώρα, τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 12α, 12 αλφα, 12 τροπολογια Δεν θα τη διαβάσω γιατί είναι μεγάλη τροπολογία, αν συμφωνείτε κι εσείς. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η παράγραφος 16, η τροπολογία 14, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 16, τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 16α, τροπολογία 16, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 17, τροπολογία 17, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, Απορρίπτεται η παράγραφος 17, τροπολογία 18, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 17α, ε, τροπολογία 19, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 18, η τροπολογία 21, υπέρ, κατά, Μισό λεπτό, καλύτερα ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. 14-12 εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην ε, τροπολογία 20 του κυρίου Ντάνιελ Φρόντ. Α, καταπίπτει. Καταπίπτει, Άρα πάμε στην 22 και τη 18α, ε, η τροπολογία 22, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε συνολικά ονομαστική ψηφορία για το σύνολο του ψηφίσματος ως τροποποιήθηκε. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Με 24, Λοιπόν, 24 υπέρ μία ε, αποχή και δύο κατά εγκρίνεται το ψήφισμα. Ε, Χαίρομαι πάρα πολύ που με βοηθήσατε ε, στο να πάρω το βάπτισμα του πυρός ε, στις ψηφορίες. Ήταν η πρώτη μου δηλαδή. Πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 6. Απαλλαγές για το Γενικό Προεπλογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018. Και θα ξεκινήσουμε τώρα συζητήσεις ή αν θέλετε ερωτήσεις προς τους ε, γενικούς ε, διευθυντές και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά Τους χαιρετίζω όλους, συλλήβδιν. Και θα δούμε τώρα ποιος, ε, πώς είναι εδώ. Έξι είναι. Έξι χαιρέτησα. Ε, λοιπόν, ε, να χαιρετήσω τον κύριο Πλέβα, Γενικός Διευθυντής ε, για την Γεωργία και την Γεωργική Ανάπτυξη, τον κύριο Μάρκ Λεμέτ, Γενικό Διευθυντή για θέματα περιφερειακή και χωροταξική πολιτική, Γιώστ Κόρτε, Γενικό Διευθυντή για απασχόληση, κοινωνικέ υποθέσει και μη αποκλεισμού, Γενική Διευθύντρια Μισού για τη μετανάστευση ε, α, η κυρία Μίχου, με συγχωρείτε. Η κυρία Παρασκευή Μίχου, Γενική Διευθύντρια για θέματα μετανάστευση και εσωτερικών υποθέσεων. Και τέλος, τελευταίο, ο κύριο Κιον Ντούνς, ε, στη συνεδρίαση των συντονιστών είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι οι γενικοί διευθυντές που ανέφερα θα κάνουν μία μικρή εισαγωγή και μετά υπάρχει δυνατότητα να τεθούν ερωτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλου στον κύριο Ζαν Ρικ Πακέ, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής για θέματα έρευνας και καινοτομίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτέ. Με μεγάλη μου χαρά είμαι εδώ τώρα στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού για να σα δώσω μια γενική έποψη για το τι έγινε φέτο, αλλά επίση να σα δώσω και μια ιδέα για την πολιτική μα, για την καινοτομία, για τα αποτελέσματα που αποσπάσαμε και το βασικό μήνυμα για αυτή την ετήσια έκθεση ε, αφορά την γενική μα διεύθυνση για καινοτομία και έρευνα και έχουμε επίσης και τις άλλες γενικές διευθύνσεις και τις άλλες υπηρεσίες που υλοποιούν αυτά τα προγράμματα και βέβαια πρέπει πολύ σοβαρά τις ε, οικονομικές τους υποχρεώσεις να είστε βέβαιοι ότι εμείς θα εξασφαλίσουμε ότι έτσι και θα συνεχιστεί. Τώρα για να δούμε τι γίνεται με την ετήσια έκθεση. Ε, ξέρετε το τι έγινε με τους ε, στόχους, τι έγινε με τις επιδόσεις, τι έγινε με τον εσωτερικό έλεγχο και τώρα έχουμε τα δύο προγραμματά πλαίσια στα πλαίσια του ε, προγράμματος πλαίσιου 7 ε, σε σχέση με το Horizon 2020, τη νέα πρόταση, να δούμε αν θα υπάρξει διοργανική συμφωνία, αλλά βέβαια έχει ξεκινήσει και η υπόθεση της υλοποίηση εν ώψη του 2021. Ε, έχουμε δύο επιφυλάξεις σε αυτή την έκθεση που είναι γνωστές, δεν είναι κάτι το καινούργιο, πριν και στην προηγούμενη έκθεση, αφορά την τις πληρωμές και ανακτήσεις ε, πληρωμών σύμφωνα με το πρόγραμμα πλαίσιο. Ε, πρόκειται για κάτι που μας κληροδοτήθηκε από το πρόγραμμα πλαίσιο και επίσης το ποστό σφάλματος είναι λίγο παραπάνω το 2%. Οπότε σήμερα με την πρακτική της Επιτροπής ε, παγίως έχουμε τις σχετικές επιφυλάξεις. Οπότε Τέλειωσε ο εσωτερικός οικονομικός ε, έλεγχος, δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα και για το μέλλον τώρα προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με το Ορίζον 2020 και τον οικονομικό έλεγχο και αντιλήσαμε συμπεράσματα από το πρόγραμμα πλαίσιο 7 και από την αρχή του Ορίζον 2020 προσπαθήσαμε να έχουμε σημαντικά μέτρα απλούστευσης και τα επέδωσαν τους πρώτους καρπούς και μετά τον οικονομικό έλεγχο και μετά αυτό το ποσοστό σφάλματος και θα προσέξετε ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω. Κύριε Γενικέ Διευθύντα, οι διερμηνείς σας παρακαλούν ή δυνατόν λίγο πιο αργά γιατί ε, οι διερμηνείς φοβούνται πάρα πολύ ότι θα χάσουν σημαντικά πράγματα από την ομιλία σας γιατί μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, ναι, συμπαθάτε με λίγο διευθυντής Οπότε τώρα προχωρούμε, κάνουμε προσπάθειά μας για το 2020 και τώρα συνεχίζεται για τα καλά η διαδικασία του ελέγχου. Η προ... Το πρώτο θετική καρπή, οι θετικέ συνέπειες για ε, το τι ήδη έχουμε μάθει και όλα αυτά ισχύουν τώρα για την αρχή του νέου προγράμματος ορίζον όσον αφορά τον ενίο συντελεστή, το μοναδιαίο κόστος, ε, ιδίω όσον αφορά το έμεσε δαπάνε και όλα αυτά τα απλουστευτικά μέτρα τα συζητήσαμε μέσα στο παρελθόν αλλά και με το ελεγκτικό συνέδριο. Οπότε τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν θετικέ επιπτώσει στο ποσοστό σφάλματο για το ορίζον 2020 και το σφάλμα συρρυκνώνεται. Βέβαια δεν μπορούμε να σταυρώσουμε τα χέρια. Ε, αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα με τον οικονομικό λόγο αλλά τέλος πάντων η τάση είναι θετική και θα είδατε ότι για το 2020 δεν έχουμε επιφυλάξει όσον αφορά την ετησία έκθεση και το εκτιμόμενο προς το λάθος πάει εκεί που θέλαμε 2 με 5% ακριβώς αυτό που είχε εξαγγελθεί ε, από και με την πρόταση της Κομισιόν το 2020 τώρα είναι το πρώτο πρόγραμμα ε, το ερευνητικό με τέτοια αποτελέσματα σε συνδυασμό με την δέσμευσή μας να μειωθεί το σφάλμα. Είπαμε την προσπάθεια απλούστευσης και ε, είμαστε περήφανοι ε, και εμεί και το επιτελείο μας και η προκάτοχή μας ότι το ελεγκτικό συνέδριο το επιβεβαίωσε ότι τα μέτρα αυτά είχαν θετικές συνέπειες επίσης όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι οι εταίροι μας το ανεγνώρισαν αυτό, όλοι όσοι το πρόγραμμα και οπότε αυτή η έκθεση ε, που γνωρίζει αυτή την θετική αξιολόγηση και επίσης η ε, συστάση είναι να συνεχιστεί η απλούστευση και όσον αφορά τον, ε, την προπαρασκευή του Horizon Ευρώπη αλλά και για την υλοποίηση αυτού. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να εξασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα θα υλοποιείται αποτελεσματικά, θα απλουστεύεται που είναι καλό για τους δικαιούχους αλλά και για την δημοσιονομική επιτυχία της υλοποίησης. Η επιτυχία του 2020 βέβαια δεν αφορά μόνο την απλούστευση και τους κανόνες υλοποίησης. Να σας πω κάποια στοιχεία για τις συνέπειες του προγράμματος γιατί ήδη την πρώτη τετραετία του βοήθησε πάνω από 300.000 ερευνητάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 17 νομπελίστες που χρηματοδοτήθηκαν από το 2020. Δεν λέω ότι έτσι γίνανε νομπελίστες, θα γίνει και αυτό, αλλά πάντως υποστήριξαμε τους καλύτερους όσον αφορά τα προγράμματα, τα, τα projects και βέβαια πάρα πολλοί πρωταγωνιστές της καινοτομίας στην Ευρώπη Οπότε τώρα ε, ε, εστιαζόμαστε στην έρευνα που πηγάζει από την υγιή περιέργεια και τέλος πάντων το πρόγραμμα ε, επικεντρώνεται στα προβλήματα της κοινωνίας και προσπαθούμε να αποσπάσουμε αποτελέσματα και για τις νέες τεχνολογίες του μέλλοντος. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο πρέπει και μπορούμε να κάνουμε περισσότερο όσον αφορά τις ευρεσιτεχνίες. Έχουμε ήδη δώσει 500 και άλλες 800 ε, εκκρεμούν η έγκρισή τους, οπότε να η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων ε, σε μεγάλη κλίμακα και ελπίζω να κάνουμε ακόμα περισσότερα κατά την υπόλοιπη διαδρομή του προγράμματος. Επίσης, προσπαθούμε με τα ερευνητικά προγράμματα στην Ευρώπη να εστιαστούμε εκεί που υπάρχει προστιθεμένη αξία και αυτό βέβαια πρώτα-πρώτα αναδύεται ε, σε σχέση με τη βιομηχανία, με την προσπάθεια των κρατών μελών, γιατί τα κρατη έχουν τη μέρα του λέοντος, εμείς δίνουμε το 8%. Ε, αλλά ε, υπάρχει δομικό αποτέλεσμα του Horizon. Θέμα να βρεθεί η κρίσιμη μάζα, να βρεθεί η προσθέμενη αξία, αλλά επίσης να υπάρχει και η συνεργασία ε, για η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και διαφόρων φορέων εκεί βασίζεται η ευρωπαϊκή έρευνα και από εκεί προκύπτει η ποιότητα των αποτελεσμάτων και όλο ένα και περισσότερο προσπαθούμε να δούμε σε τρίτο πλάνο για την προστιμένη αξία να βοηθήσουμε τα κρατη για τα γεωπροβλήματα της κοινωνίας και το ορακό πρόγραμμα δεν είναι προστιμένη αξία ότι πολλές φορές ε, αφορά πάρα πολλέ ε, πολιτικές, πάρα πολλέ επιστήμες, κάτι το οποίο δεν το κάνουν τα εθνικά προγράμματα. Επίσης είναι πάρα πολύ ευέλικτο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να βοηθάει για κάποιες λύσεις όσον αφορά τις ε, πολιτικές τη Ευρώπη, τεχνολογία, κοινωνικά θέματα, επιστήμη και τεκμηρίωση των πολιτικών. Οπότε σκεφτόμαστε στο πώ θα βοηθήσουμε όλα αυτά, οπότε βοηθούμε και τη χάραξη πολιτικών. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, πρόεδρο. Ναι, ναι, ναι, κλείνω, κλείνω, πρόεδρε. Το ορίζον 2020 έχετε βελτίωση και αυτό που τώρα να κάνουμε με το Οριζόν Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να επεξεργαστούμε το τι γίνεται με την υπερβολική ζήτηση γιατί πάρα πάρα πολλοί θέλουν να μπουν. Ε, αυτή είναι η μακρογωνία τάση και αυτό εξηγείται γιατί το πρόγραμμα είναι επιτυχημένο επίσης ε, γιατί οι περισσότεροι ποντάρουν στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διαδικασία της αξιολόγησης πρόκειται όλα αυτά να τα λάβει υπόψη. Υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση, γι' αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και θεμητή. Πώς δηλαδή το πρόγραμμα μπορεί καλύτερα να βοηθήσει τους ερευνητάς σε όλα τα κρατή-μέλη. Ε, βέβαια πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο για την καινοτομία. Και έχουμε το σχετικό συμβούλιο, πρόταση της Κομισιόν του κυρίου Μουέντας και αυτό θα μπει επίσης ε, στην διαδρομή του ορίζοντα 2020. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Και ε, ευχαριστώ να απαντήσουμε ερωτήσεις των μελών. Σας ευχαριστούμε κύριε Γενική Διευθυντά. Επειδή είμαι εισηγήτρια, παρότι δεν νύθιστε ο πρόεδρο να λαμβάνει προς το λόγο, εγώ θα ξεκινήσω με τι ερωτήσει, αν με επιτρέπετε. Ήδη αναφερθήκατε σε κάτι και εσείς ο ίδιος, ε, δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα ε, μεμονωμένα ε, που είναι καλά, 7 με 20 αλλά έχει ξεπεραστεί ο, ο στόχος και θα πρέπει να δούμε την ισότητα, την, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ισότιμο. Ε, και πολλές φορές ε, η διαφορά μπορεί να είναι 0,1-0,2 είναι λίγο αυθαίρετο δηλαδή, ε, αυθαίρετος τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να τα επιλύσουμε και δεν νομίζω ότι υπάρχει και η κατάλληλη ίσως ενημέρωση αναφορά από τους υπουργού έρευνας, υπουργού οικονομικών. Ε, το ερώτημά μου είναι η συνεργασία με τις εθνικές διοικητικές δομές, αρχές, πώς ε, συντονίζεται, πώς ε, λειτουργεί. Υπάρχει ένα είδος ανταγωνισμού ενδεχομένως ε, στο έργο των κρατικών αρχών. Έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο, το αναφέρετε κι εσείς, ότι ήδη έχει υπάρξει κάποια πλούστευση και νομίζω ότι το αναφέρει αυτό ρητός και στην έκθεση του το ελεγκτικό συνέδριο όμως ε, σε ό,τι αφορά τα πανεπιστήμια που δεν ε, είναι ίσως ε, το ίδιο πεπειραμένα κέντρα αριστείας δυσκολεύονται ενδεχομένω να καταθέσουν τις αιτήσει. Πόσο λοιπόν συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και σε ό,τι αφορά τώρα το πρόγραμμα πλαίσιο το έβδομο, ε, το οποίο αφού κλείσει πρέπει να αξιολογηθεί βεβαίως. Ε, υπάρχει αυτό το υπόλοιπο προς εκαθάριση το οποίο έχετε αναφέρει 57,3. Όμως από τη στιγμή που έχει κλείσει αυτό το πρόγραμμα πώς, ποιο είναι το υπόλοιπο, το πραγματικό προς εκαθάριση που είναι διαθέσιμο και ε, εγώ ολοκλήρωσα, αυτό δώσω τώρα στους Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Με τη σειρά να απαντήσω ε, εγώ. Πράγματι είναι πρόβλημα αυτό που είπατε ε, για τις ερευνητικές κοινότητες ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το κόστος προετοιμασίας μιας πρότασης είναι σημαντικό. Η πραγματική απογοήτευση έγκυται όμως στο ποσοστό επιτυχίας 11, ε, ε, μήπως και 3 και 4 μπορεί να είναι και πολύ χαμηλότερο, που δεν είναι θετικό. Και αυτό που μας απογοητεύει είναι ότι αυτό το ποσοστό επιτυχίας 25% ε, ε, αφορά προτάσεις ποιοτικέ, ποιοτικά, ε, το είπατε και εσείς, προγράμματα για τα οποία όμως δεν υπάρχει προϋπολισμός. Και πραγματικά είναι δύσκολο αυτό να το δούμε, γιατί φυσικά και εξαρτώμεθα από την κινητοποίηση στην Ευρώπη, η ποιότητα των προγραμμάτων λοιπόν είναι θέμα. Και σε πολλά κράτη-μέλη οι πόροι για την έρευνα και την καινοτομία δεν είναι πάντοτε προτεραιότητα ε, και δεν... Ε, μπορώ να πω ότι πάντοτε τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Πολλές φορές είμαστε θύματα της επιτυχίας μας, αν θέλετε. Τα συζητούμε και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Τονίζουμε την ανάγκη να γίνουν εθνικέ επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει η συζήτηση, όλη η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και ήδη βλέπουμε βελτιώσει σε πολλού τομεί. Τώρα, πώ θα το αντιμετωπίσουμε. Αφενό, ε, με τέτοιου είδου πιέσει προ το σύστημα, η έννοια τη διαφάνεια, η έννοια τη δικαιοσύνη, ούτω ή άλλω δηλαδή είναι σημαντικά, αλλά εδώ είναι ακόμα πιο σημαντικά θέματα και το είπατε κι εσεί, η χρηματοδότηση μπορεί να βασίσει το 0102 σε ένα τέτοιο περιθώριο διαφοράς. Και νομίζω οι εξολογήσεις ε, χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό, διαφάνεια, οι διαδικασίες ε, τρέπουν επίσης ε, την επανόρθωση, την εξέταση των αποτελεσμάτων και πολλές φορές αξιοποιούν την δυνατότητα αυτή οι εκτελεστικοί οργανισμοί που κάνουν το, την αξιολόγηση ε, έχουν αναλάβει αυτή τη δουλειά. Και τώρα επειδή προετοιμαζόμαστε και για το Horizon Europe, αυτά τα συζητούμε με τους εταίρους μας για να δούμε πώς μπορεί να συνεχιστεί ε, πλήρως αξιόπιστα και διαφανώς αυτή η διαδικασία αξιολόγησης. Νομίζω ότι η έννοια της ε, μεροληψίας που βασίζεται στη φήμη, reputational bias. Μπορεί να το έχετε ακούσει αυτό. Το γνωρίζουμε. Η λύση δεν έγκυται στον προπολογισμό, δεν θα είναι τετραπλάσιος ο προπολογισμό στο ορίζον Ευρώπη, άρα δεν θα λυθεί το πρόβλημα έτσι. Στα προγράμματα εργασίας μπορούμε να βρούμε λύσεις, δηλαδή εστιάζοντας πολύ καλύτερα ε, ώστε να καθοδηγούνται οι ερευνητές και να είναι λιγότερες οι περιπτώσεις που καταθέτουν πολλές προτάσεις που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα και στο επίπεδο αξιολόγηση. Και έχουμε και τα πιλωτικά στις ε, δύο φάσεις της αξιολόγησης. Γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα στην πρώτη φάση και πάνε λιγότερες, λιγότερες προτάσεις στη δεύτερη φάση. Ελπίζουμε τόσο πάντων να το λύσουμε το πρόβλημα, αλλά είναι καλό το πρόγραμμα σίγουρα και υπάρχουν υψηλέ προσδοκίες από τους ερευνητές και ανάγκες για τους κανόνες που είναι πολύπλοκοι. Αυτό εν μέρει οφείλεται στο ότι η αρχή είναι η επιστροφή του επιλέξιμου κόστους. Γι' αυτό απαιτούνται σαφείς οδηγίες και σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση και την εφαρμογή. για τους νέους νοησερχόμενους αυτό είναι μια πρόκληση. Οι μισοί συμμετέχοντες στο νέο πρόγραμμα είναι νέοι και είναι μεγάλη πρόκληση. Για να μπορούν όλοι δηλαδή στο, στην Ευρώπη να κατανοήσουν ε, το πρόγραμμα. Όταν κάποιο είναι νέος δεν πρέπει δηλαδή να έχει περαιτέρω εμπόδια για να κατανοήσει τις διαδικασίες. Υπάρχουν και τα δίκτυα των εθνικών συνδέσμων. Αλλά υπάρχουν και ομάδες της Κομισιόν και των εκτελεστικών οργανισμών επιτόπου στα κράτη-μέλη πηγαίνουν και βοηθούν τους δικαιούχους να καταλάβουν τους κανόνες του προγράμματος. Και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτό. On the, um, on, uh, FP... Για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, 100 προγράμματα παραμένουν ανοιχτά σήμερα. Θα έχουν κλείσει μάλλον μέχρι τα τέλη του 20. Άρα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την επιτόπερ το βλέπουμε στην ακτού το τέλος του προγράμματος. Αλλά μάλλον θα περάσουν λίγα χρόνια ακόμα μέχρι τυπικά και επίσημα να κλείσουν όλα τα προγράμματα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του ελέγχου. Άρα έχουμε κάποια χρονάκια μπροστά μας πριν βάλουμε πίσω μας το 7. Ε, δεν το κατάλαβα αυτό που είπε το ότι είναι στο τούνελ, το βλέπουμε, ε, ότι όπου να είναι κλείνει, αλλά έχουμε κάποια χρόνια ακόμα. Δηλαδή τι, καθυστερεί ένα χρόνος, δύο χρόνια. Πρόεδρος, όχι, δεν καθυστερεί. Υπάρχουν προγράμματα 100% ανοιχτά που θα κλείσουν. και τα 100, μάλλον ε, προγράμματα που είναι ανοιχτά, δεν θα κλείσουν όλα. Ε, αλλά ε, μέχρι τότε. Σιγά σιγά θα κλείνουν, αλλά μέχρι το τέλος του 20 θα έχουν κλείσει όλα, τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω. Επελέγησαν το 13. Το 13 και το 14 έγιναν αναθέσεις. Για το ραλ, για το υπόλοιπο προσεκαθάριση που είπατε, δεν τα θυμάμαι τα νούμερα, θα τα δω και θα σας τα στείλω. Το υπόλοιπο προς εκαθάριση, σε ό,τι εξ όσων γνωρίζω, είναι υπό έλεγχο. Και νομίζω ότι αυτό που λέω είναι βέβαιο. Αρκετά χρόνια κρατάει η λειτουργία και των προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, τις χρησιμοποιούμε τώρα. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα ε, μια μικρή πίεση της τάξης του 1,5% όταν δεν έχουμε ε, όλες τις αιτήσει εντεγκέρως. Ε, αλλά είναι υποέλεγχο η κατάσταση και θα σας δώσω βέβαια και τα στοιχεία όταν τα βρω. Η Σκιώδης παρακαλώ τώρα. Πένκοβα και μετά σας στέλνω. I don't have a question. Εγώ δεν έχω ερώτηση. Εσείς έχετε, δύο σας θέλει. Ναι, κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, εγώ έχω μια ερώτηση προς εσάς. Όταν έχουμε ένα εγκάρσιο ερώτημα που αφορά όλους τους γενικούς διευθυντές, το θέτουμε, περιμένω να απαντάνε όλοι με τη σειρά τους. Ναι, ή αλλιώς το ξαναθέτει το ερώτημα. Βεβαίως, βεβαίως, μάλιστα. Λοιπόν, το πρώτο μου ερώτημα είναι τέτοιου είδους, απευθύνεται σε όλους δηλαδή τους γενικούς διευθυντές, ε, και βασίζεται και στην έκθεση απαλλαγής για το 17.000, ε, συγγνώμη, σημείο 220. Το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη για το ότι τις εκθέσεις πεπραγμένων δεν αναφέρουν στοιχεία για την ποιότητα των στοιχείων που από τις απόδοση των επιδόσεων. Δηλαδή, εγκρίνοντα την ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τι επιδόσει, το Σώμα των Επιτρόπων αναλαμβάνει την ε, πολιτική, τη γενική πολιτική ευθύνη για τη χρηματοοικονομική διαχείριση του προπολογισμού τη Ένωση, αλλά όχι σε ό,τι αφορά τι πληροφορίε για τι επιδόσει και τα αποτελέσματα. Αυτά τα λέει η έκθεση απαλλαγή του 17 και επανέρχομαι σε αυτά γιατί θα ήθελα να μου πούν οι γενικοί διευθυντέ ποια είναι η άποψή του γι' αυτό. Δηλαδή η πολιτική ευθύνη περιλαμβάνει την ευθύνη των γενικών ε, ε, διευθυντών ή είναι κάτι διακριτό. Έχετε λάβει μέτρα για να βελτιώσετε το γενικό σύστημα μέτρησης των επιδόσεων με δείκτες αποτελεσμάτων σε επίπεδο project, έργων για να από, εξακριβωθεί κατά πόσον οι στόχοι πληρούνται από τα προγράμματα. Αυτό είναι ένα γενικό ερώτημα προς όλους τους διευθυντές και σε ό,τι αφορά τη ερευνα έρευνα. Είχα δύο-τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτη αφορά την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Υπάρχουν κριτήρια για την ανάθωση προπολογισμού στον όρο του 2020 και ξέρω ότι γίνονται πολλές προσπάθειες. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής, θα ήθελα κάποιε επεξηγήσεις το gender mainstreaming βοηθάει ώστε να έχουν οι γυναίκες και οι άντρες τις ίδιες ακριβώς ευκαιρίες πρόσβαση χρηματοδότηση. Γιατί στην έκθεση για τα τέλη του 2018 ε, ήταν 21.000 και κάτι οι Και μια ερώτηση. Επειδή με ενδιαφέρουν οι ΜΜΕ, σήμερα πώς αξιολογούμε το επίπεδο συμμετοχής ΜΜΕ ψηλών. στο πρόγραμμα 20, στο 2020 και στα συγκεκριμένα σκέλη που τις αφορούν. Si vous le permettez, Madame la Présidente, Monsieur Châtel, pour la question relative à la performance, Σχετικά με τις επιδόσεις μας, ναι, πρέπει να είναι εγκάρσια, οριζόντια η απάντηση, γιατί πρόκειται για θέση του σώματος των επιτρόπων. Οπότε να μην σας τα πω εγώ, αλλά σας τονίζω ότι ε, στην έκθεση είναι πάρα πολύ σαφείς οι επιδόσεις μας είναι άμεση η διαχείριση της έρευνας από την Κομισιόν, από τις ε, περιφερειακές υπηρεσίες, από τη Γενική Διεύθυνση και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Βεβαίω και με στη θέση σας να τα δούμε στις λεπτομέρειες του τα θέματα, αγαπητέ βουλευτά. όσον αφορά την ανισότητα των φύλων, Υπάρχει Επιτροπή Αξιολόγησης και οι εμπειρογνώμονες όπου θα πρέπει να πριτανεύει αυτή η ισότητα των φίλων όσο είναι δυνατόν. Εμείς το προσέχουμε αυτό. Να μην υπάρχει προκατάληψη στην επιλογή. Για το αποτέλεσμα πάντως δεν υπάρχει κριτήριο γιατί τα προγράμματα και τα ε, ερευνητικά προγράμματα ε, κατανέμονται με βάση την αριστεία. Και οπότε θεωρούμε ότι τα πράγματα πάνε καλά στην Ευρώπη. Πάντως 50% από τους νέους ερευνητές, από αυτούς που έχουν διδακτορικό, 48% συγκεκριμένα είναι γυναίκες, δεν πάνε άσχημα τα Από την άλλη μεριά, όσον αφορά τους επικεφαλείς των ερευνητικών κέντρων εκεί έχουμε πιο χαμηλές επιδόσεις 25 με 30% Επομένως είναι υποχρέωση, είναι μια φιλοδοξία για τα κρατημέλη να διορθώσουν τα πράγματα, οπότε θα πρέπει και τα προγράμματα να βοηθήσουν όσο γίνεται τώρα για τις ΜΜΕ. Αν δεν σας απάντησα για τις υποτροφίες. Κιουρί, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Να τα δω όλα μαζί και να τα δούμε στο λεπτομέρειες μαζί. Οπότε για τις ΜΜΕ συνδέονται με την υπόθεση της έρευνας, συμμετέχουν σε πολλά προγράμματα για κοινωνικά προβλήματα, για ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Οπότε βοηθάμε για την καινοτομία και ο στόχος είναι το 20% για τα σημερινά προγράμματα. Πολύ ωραία. συνάδελφος Βιόλα Φων Κάμον. Και εγώ θα μιλήσω σήμερα γερμανικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισήγηση. Και όσον αφορά τις ε, ερωτήσεις ε, των προλαλισάντων, συμφωνώ και εγώ αυτά τα οποία άκουσα από γερμανικά ερευνητικά ιδρύματα ή αν θέλετε από διάφορους επιστήμονες είναι ότι η πρόσβαση σε ερευνητικά κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' ουσίαν σημαίνει μια μεγάλη επένδυση. Δηλαδή ένα ερευνητικό ίδρυμα, μια μικρή νεοφύση επιχείρηση, ένα πανεπιστήμιο, όλοι αυτοί πρέπει πρώτα να προσλάβουν προσωπικό και μετά να ζητήσουν τα ερευνητικά κονδύλια. Είχα ακούσει λοιπόν ότι τελικά από τις αιτήσει ε, εγκρίνεται περίπου το 3%. Άρα το να μην εγκριθεί ένα αίτημα, αυτό είναι πολύ πιθανό και εκεί ε, χάνονται πολλά κονδύλια. Εμένα αυτό που μου λένε είναι ότι υπάρχει μία αναντιστοιχία. Δηλαδή έχουμε επαγγελματικά επιστημονικά προγράμματα όμως, από τη μια πλευρά, από την άλλη όμως δεν είναι απαραίτητα οι καλύτεροι ερευνητές και τα καλύτερα πανεπιστήμια τα οποία ε, εμείς στηρίζουμε για τα μελλοντικά μας προγράμματα. Ως εκ τούτου θα πρέπει στο επόμενο πρόγραμμά μας, το Horizon Europe, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Και από τη μία δεν θα πρέπει να υπάρχουν υπερβολικές, υπερβολικά αιτήματα τα οποία να απορρίπτονται. Από την άλλη όμως ε, να γνωρίζουν μικρά ιδρύματα και μικροί ερευνητέ ότι μπορούν και αυτοί να χρηματοδοτηθούν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όσον αφορά το θέμα, τη διάσταση των δύο φύλων, ε, πράγματι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να το προσέξουμε πολύ περισσότερο στο επόμενο ερευνητικό πλαίσιο. Έχω όμω μια τελείω διαφορετική ερώτηση και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να τοποθετηθείτε από αυτού ή αν θα μου απαντήσετε γραπτά. Άκουσα δηλαδή ότι έχουμε μία μεγάλη ε, κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας και πέρυσι η εταιρεία αυτή είχε περίπου 17 προγράμματα που εφάρμοσε και με τη γενική σας διεύθυνση, γενικότερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, όμως ε, αποδείχτηκε ότι τα προγράμματα αυτά τα στήριξε και το κυβερ... κινέζικο κράτος τα οποία κατ' ουσίαν ε, κονδύλια θα έπρεπε να επιστραφούν από τις ε, κινέζικες επιχειρήσεις. Βεβαίως ε, αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο γιατί εμείς δυστυχώς πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά στα κινέζικα και κάπου δεν τα καταφέρνουμε. Εγώ ερωτώ συγκεκριμένα, εσείς έχετε ακούσει τίποτα γι' αυτό, κάνατε κάτι απευθυνθήκατε στην Όλαφ για τη τελική ανάλυση πρόκειται για κάποια εκατομμύρια και για μένα αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι είναι θέμα αρχής. Θα το αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι ή τι θα κάνουμε. Ε, να πω κάτι που αφορά στις αξιολογήσεις και στον ρόλο που είναι πράγματι πολύ σημαντικό στο ρόλο που παίζουν οι σύμβουλοι για να προετοιμάσουν τα προγράμματα. Και όταν εφαρμόζονται τα προγράμματα, πράγματι μερικές φορές υπάρχει υποστήριξη, αλλά η έρευνα ε, θα πρέπει να γίνεται από τους ίδιους ερευνητές. Αυτό είναι απόλυτα σαφές και πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι σύμβουλοι ε, πολλές φορές ε, πράγματι είναι εκείνοι που τελικά υποβάλλουν δυστυχώς προτάσεις. Όλα αυτά τα εξετάζουμε, ε, κοιτάμε να δούμε πώς θα αλλάξουμε το θέμα, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να, γίνεται, να έχουμε δύο φάσεις. Η δεύτερη φάση να γίνεται εδώ με συνέντευξη στις Το κάναμε αυτό και είδαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Βλέπουμε, ας πούμε, τον ερευνητή ε, μπροστά σου και ξέρει να στηρίξει την πρότασή του. Υπάρχει και κάτι άλλο. Ε, υπάρχει πολλές φορές και μια ομάδα ερευνητών που είναι εξαιρετική ε, και αυτοί θα πρέπει να έχουν μια ευκαιρία. Το εξετάζουμε για να δούμε πώς μπορούν να βελτιωθούν όλα αυτά. Ε, κατά τα άλλα γνωρίζουμε πολύ καλά περί τίνος πρόκειται, τι διακυβεύεται γιατί είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πολλές γενικές διευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το στήσιμο των προγραμμάτων θα περάσουμε και στον έλεγχο για να δούμε λιγάκι τι θα γίνει με τις διάφορες ενησυχίες. Εντάξει, δεν θα απαντήσω εγώ εκ μέρους της Όλαφ, αλλά όσον αφορά την έρευνα τουλάχιστον από πλευράς ε, ερευνητικής κοινότητας, πρέπει να σου πω ότι εμείς το ψάχνουμε. Πολύ ωραία. Ο συνάδελφος Φλένιγκαν δεν είναι εδώ. Η κυρία Κρετού, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο ρόλος μας ως Ευρωβουλευτών είναι να ασκούμε κριτική, αλλά εγώ, ξέρετε, ζήτησα το λόγο για να πω και ένα ευχαριστώ για την πολύ καλή επαφή που έχουμε με τους ε, Γενικούς Διευθυντές της Έρευνας και της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Από το 2014 ήδη έχουμε προσπαθήσει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη κονδυλίων για την έρευνα και την καινοτομία. Και ε, έχουμε αυτό που αποκαλούμε σφραγίδα της αριστείας, ε, λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια, τελικά προγράμματα που δεν μπορούν να, ε, να χρηματοδοτηθούν από το Horizon 2020 να έρχονται από το ERDF. Αλλά στον επόμενο κανονισμό ε, θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο το πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στο ERDF το Horizon 2020, το Erasmus Plus, ε, για να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα στην έρευνα και ίσως ε, να βρούμε και έναν τρόπο να σκίσουμε πίεση στα κράτη-μέλη να χορηγούν περισσότερα κονδύλια στην ε, έρευνα και την καινοτομία γιατί αυτά τα δύο στοιχεία είναι η κινητήρια δύναμη κάθε κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έχετε απόλυτα δίκιο ότι η συνεργασία ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού είναι πολύ σημαντική. Εσείς ήσασταν πρωτοπόροι, συνεδριάσατε τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Horizon 2020 και η σφραγίδα της αριστείας, το Seal of Excellence, είναι κάτι ε, που πέτυχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τώρα εμείς ε, εξορθολογίζουμε το μέτρο για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία όσον αφορά τα κρατικά κονδύλια, οποτεδήποτε δηλαδή ένα κράτος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει αυτή την σφραγίδα της ε, αριστείας. Ε, να γίνεται καλύτερη χρήση αυτής της δυνατότητας. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν συνέργειες ε, περισσότερο από ό,τι συμβαίνει σήμερα και οι δύο γενικές ε, διευθύνσεις συνεργάζονται με το Κοινοβούλιο και με άλλους εμπειρογνώμονες, τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσουν ότι οι κανόνες που αφορούν τα διαφορετικά ταμεία αλλά και μας ε, να μπορούν να εφαρμόζονται στο μέγιστο βαθμό. Γίνεται πάρα πολύ δουλειά αλλά ε, ακόμα υπολείπονται πολλά ε, στην διαδικασία της αναπόφασης για το Horizon 2020 και για άλλα. Το Κοινοβούλιο μπορεί να μας βοηθήσει να επιτύχουμε το νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να έχουμε συνέργειες όσο το δυνατόν περισσότερο και βεβαίως εναπόκειται στην Κομισιόν και στους αρμόδιους να ε, βοηθήσουν έτσι ώστε όσοι θέλουν να μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των συνεργειών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό καθήκον, γιατί έχουμε ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία σε επίπεδο πανεπιστημίων δεν αποφελούνται σχεδόν καθόλου. Και έχουμε επίσης και το πρόβλημα ότι ε, μέχρι τώρα μπορούμε να προάγουμε την αριστεία, αλλά όχι ε, να ε, βοηθήσουμε ώστε να συνεργάζονται πανεπιστήμια στο μεσαίο επίπεδο. Δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί με τις οικονομικές μας δυνατότητες. Θα ήταν όμως ένα στόχος αυτό για να γινόμαστε ακόμα πιο άριστοι. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε και αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις θα απευθυνθούμε σε εσά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, πάω στον ε, επόμενο ε, Γενικό Διευθυντή. Περνάμε στην Γεωργία. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις δικές σας τις απόψεις. Madam Chair, honorable members, thank you for... Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω τις σχέση και, πραγμένων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, της Διάγκρη. Θέλω να σας δώσω μια πραγματική εικόνα της κίνησης της πολιτικής και του τι κάνουμε στην Άγκρη Το 2018. ήταν μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά με πολλά επιτεύγματα. Το νέο οργανικό οργανισμό του Ιουνίου του 2018 που ορίζει τα θεμελία της περαιτέρω επέκτασης για την εναρμόνιση των, μάλλον με την εναρμόνιση των κανόν και τη δημιουργία ενισότιμου πεδίου ανταγωνισμού το σύστημα των άμεσων πληρωμών και το παρασύνδεσμα καλύπτει το 100% των ε, χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων. Οδηγία για αθέμητες εμπορικές πρακτικές, UTPs. που συμφωνήθηκε το τέλος του 18 θα προστατεύει τους πλέον αδύναμους και θα οδηγήσει σε επανεξισορρόπηση των δυνάμεων στην αγορά της αλυσίδας τροφίμων. Το 18 είχαν περίπου 7 εκατομμύρια δικαιούχους που έλαβαν στήριξη εισοδήματος ε, ή επενδύσεις για τις εκμεταλλεύσεις τους ή για πρακτικές φιλοπεριβαλλοντικές. Λίγα μόνο παραδείγματα σας δίνω. Κατάσταση της αγοράς. Σημείωσε περαιτέρω βελτίωση. Μεγαλύτερη σταθερότητα και ανάκαμψη από την κρίση. Η αιτήσια πεπραγμένων δείχνει πως ό,τι αφορά την κατανομή των άμεσων πληρωμών ε, δεν είναι τόσο άσπρο-μαύρο όπως μπορεί να το καταλαβαίνει το κοινό. Ε, υπάρχουν διακοιμάσεις. Το 72% των άμεσων πληρωμών του 18 κατεβλήθησαν σε επαγγελματικέ οικογενειακέ ε, αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 5 έω 250 εκτάρια. Περισσότερες αυτά, τα περισσότερα από αυτά τα αγροκτήματα δεν ξεπερνούν τα 20 εκτάρια όμω. Εμεί θα συνεχίσουμε να κάνουμε πιο πολλά για να υπάρχει ακόμα πιο δίκαιη κατανομή των πληρωμών για την ΚΑΠ μετά το 2020. Εκτέλεση προγραμμάτων. Είχαμε εξέλιξη στο World Bank, στην Παγκόσμια Ανάπτυξη, 48%, πάνω από 140.000 αγροκτήματα πήραν το 18 υποστήριξη για αναδιάρθρωση και εξυγχρονισμό. Το 40% επίσης των αγροτικών εκτάσεων ήταν για πήραν στήριξη για φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα και έχουμε και 106.000 νέους αγρότες που ωφελήθηκαν από τα μέτρα στήριξης. Τα νέα γεωργικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά. Τα γεωργικά προϊόντα της Ένωσης είναι ανταγωνιστικά και είμαστε κοντά στη μέση τη αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΑΓΚΡΙ έπαιξε σημαντικό ρόλο στι διαπραγματεύσει εμπορικών συμφωνιών με Ιαπωνία, Καναδά, Μεξικό. Και συνεχίζουμε να προωθούμε ενεργά την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα χώρε εταίρους. Έχουμε και διάφορες task force όπως αυτή για την Αφρική που συνέβαλε σημαντικά στην Συμμαχία Αφρικής Ένωσης, Ευρώπης μάλλον, για επενδύσεις σε θέσεις απασχόλησης. Τις η εκθέσει πεπραγμένων ορίζει και κάποιες ε, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. λείπεται των μισθών της, ε, των άλλων οικονομικών κλάδων το εισόδημα των ε, Γιώργο. Γι' αυτό και χρειάζονται άμεση υποστήριξη. συνδεσιμότητα. Υπάρχει ένα κενό στι ε, περιοχές υπαίθρου σε σχέση με την πρόσβαση σε νέας γενιάς ε, τεχνολογίες στο διαδίκτυο. Πρέπει να καλυφθεί το κενό. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές θερμοκηπιακού αερίου, θερμοκηπιακών αερίων. Υπάρχουν πιέσεις σε αέρα, νερό, έδαφος. Και σε ό,τι αφορά τη μέτρηση των επιδόσεων, πρέπει να βελτιώσουμε κάποιους δείκτες. Η Γενική μας Διεύθυνση, σας διαβεβαιώ, θα συνεχίσει να, να κάνει πάντο δυνατόν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων προς όφελος των Ευρωπαίων αγροτών και της κοινωνίας εν γέννη. Και τώρα πανέρχομαι στο οικονομικό έντος 18 και το τι πετύχαμε. Θέλω να τονίσω ότι η ΚΑΠ είναι ένα σημαντικό κομμάτι των δαπανών, 38%. Καλή διαχείριση για το 18, το 98% περίπου των δαπανών στο πλαίσιο της ΚΑΠ δεν είχε κανένα σφάλμα. Το ποσοστό σφάλματος συνολικά για την ΚΑΠ είναι 2,15%. Δηλαδή χαμηλότερο από το προηγούμενο έτος. Πολύ κοντά στο 2%. Για τις άμεσες πληρωμές για το Γεωργικό Τάμιο. 1,83% ήταν το ποσοστό σφάλματος. Κάτω από το στατιστικά σημαντικό δηλαδή όριο, το 2%. Και για το ΕΤΠΑ επίσης μείωση του ποσοστού σφάλματος. 3,2% ήταν το ποσοστό του το 18. Όμως, ο χαμέτερος ε, κίνδυνος είναι κάτι που πρέπει να τονίσουμε. Τα κράτη μέλη κάνουν προσπάθειες να αντιμετωπίσουν ε, τα αίτια σφάλματος. Εφαρμόζουμε βέβαια και καθαρές οικονομικές διορθώσεις. Άρα, συνολικές διορθωτικές ενέργειες οδήγησαν για το 18 σε ένα ποσοστό 0,25 για ανάγκη διορθώσεων. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα. Και θα συνεχίσουμε έτσι για να αντιμετωπίσουμε και τις μελλοντικέ προκλήσεις. Πρόταση για τη μετά το 2020 κοινή γεωργική πολιτική είναι η διποσυζήτηση σε επίπεδο των νομοθετών. Πρόεδρο, σας παρακαλώ αν μπορείτε να ολοκληρώσετε. στόχος της πρότασης είναι να αντιμετωπίσετε τις ανησυχίες που είχατε εκφράσει κατά το παρελθόν σε ψηφίσματά σας για την απαλλαγή, δηλαδή πιο δίκαιη ε, κατανομή των άμεσων πληρωμών, μείωση του διοικητικού άχθους, επίσης εστίαση στις επιδόσεις, περιβάλλον και νομίζω ότι θα μπορέσουμε από κοινού να δημιουργήσουμε ε, μια πιο σύγχρονη και δίκαιη κοινωνική πολιτική για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας αυτή την παρατήρηση. Και επειδή εγώ είμαι η συγγητρία, ξεκινάω με τις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι η Επιτροπή Κοντα ασχολήθηκε σε βάθος με θέματα που αφορούν τη σύγκρουση συμφερόντων ε, στην Τσεχία και στη Σλοβακία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω τι μέτρα λάβατε που να αφορούν σε αυτές τις περιπτώσεις ε, που έγιναν γνωστές, γιατί από αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα δεν ακούσαμε τίποτα. Δεύτερη ερώτηση. Εν τω μεταξύ, ε, στηρίζονται συνεταιρισμοί οι οποίοι έχουν συσταθεί έτσι ώστε να θέτουν στην αγορά διάφορα προϊόντα. Και εδώ έχουμε ακούσει κάποιες περιπτώσεις στην Πολωνία όπου ε, δεν στηριχθήκαν μόνο οι συνεταιρισμοί, αλλά αγοράστηκαν με ευρωπαϊκά χρήματα και τα δέντρα, οι μιλιές, όχι μόνο τα μήλα. Ε, και αυτό για να προσφέρονται τα προϊόντα σε ευνοϊκότερες ε, τιμές. Ε, Βεβαίω τα σχετικά έγγραφα θα σας τα χορηγήσω θα ήθελα απλά να σας επισημάνω ότι εντωμεταξύ διάφορες χώρες διαμαρτύρονται ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν άμεσα για την γεωργική παραγωγή και δεν ακολουθήθηκαν οι σχετικές διατάξεις. Κατά τα άλλα, όσον αφορά στους ενεργούς γεωργούς, τους νέους γεωργούς και, την, και τις βιολογικές καλλιέργειες. Ε, υπήρξαν κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, σχετικά με ελλείμματα που αφορούν στο σύστημα LPIS, Land Identification System, του εντοπισμού, του γεωργικού εντοπισμού, ε, τα κράτη-μέλη. Πώς ε, σκοπεύετε να το διευκρινίσετε το θέμα, γιατί ξέρετε εμείς θέλουμε τα κονδυλιά μας να φτάνουν ε, εκεί που πρέπει και όχι σε λάθος χέρια. Κατά τα άλλα, γνωρίζουμε επίσης στη Σλοβακία, αλλά εντωμεταξύ και στη Ρουμανία, περιπτώσεις όπου υπήρξε η φαρπαγή γης από μικρούς γεωργούς. Και θέλω να ρωτήσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έκανε γι' αυτό. Γιατί αυτό δεν μπορεί να επιληθεί με ένα σύστημα εντοπισμού. Βεβαίως ε, η γη και οι καλλιέργειες είναι γνωστές, αλλά αυτό που μου είπαν εμένα είναι ότι τελικά χρησιμοποιούνται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και όταν υπάρχει αυτή η παράνομη φαρπαγή γίνονται πλαστά, προκύπτουν πλαστά έγγραφα και με τον τρόπο αυτό μπορεί ο, ο, εκείνος που υφαρπά στην γη ακόμα και να ε, νομιμοποιήσει την πράξη του. Το τελευταίο μου ερώτημα όσον αφορά την εκχέρσωση λόγω πυρκαγιάς και τη Μερκοσούρ, της χώρας Μερκοσούρ. Εμείς ε, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι επειδή υπάρχουν πυρκαγιές και μετά προκύπτει εκχέρσωση γης, δεν θα πρέπει αυτό να βλάψει ε, το δικό μας τον τομέα ξυλίας. Αναφέρομαι κυρίως ε, στις χώρες Μερκοσούρ. Τώρα, για τα μήλα από την Πολωνία, σας είπα, θα σας στείλω και τα σχετικά έγγραφα. Thank uh, Πολύ σπουδές αυτές οι Ευχαριστώ. Να αρχίσουμε με αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με Τσεχία και Σλοβακία, όλες αυτές οι υποθέσεις που εφήξατε. Οπότε, το έχουμε πάρει το θέμα στην κοινή της πολύ σοβαρά. Επεμβαίνουμε διορθωτικά. Κάναμε από τον Ιανουάριο μια ερευνητική αποστολή να δούμε τι γίνεται όσον αφορά και υπήρχε επίσης συντονισμός με την DG Regio και απασχόληση για έλεγχο. Συνεχίζεται αυτή η έρευνα για να δούμε ε, πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία ε, της κατά αντιπαράθεση εξέτασης. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε πάντως τις ε, λεπτομέρειες γιατί είναι πολύ σημαντική η εμπιστευτικότητα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι αυτή η κατά αντιπαράθεση διαδικασία θα είναι στεγανή και δίκαιη. Ως ε, προπαρασκευαστικά ή μάλλον ε, μέτρα εξασφάλισης δεν εκταμιεύουμε χρήματα από τα επενδυτικά και δηλωτικά ταμεία προς εκείνες τις εταιρείε που ενέχονται άμεσα ή έμεσα με όσους θα μπορούσαν να κρυφθούν επιλήψιμοι, πρωθυπουργοί κλπ. Και με τις αρχές της ε, χώρας προσπαθούμε να δούμε τι ποσά μπορεί να είναι αυτά τα οποία έχουν σχέση με επιλήψιμους στη διαδικασία. Τώρα όσον αφορά την μη τήρηση της διαδικασίας, έχουν ληφθεί τα σωστά μέτρα, τα πιο δόκιμα για τον προϋπολογισμό, διορθωτική παρέμβαση, για το παρελθόν, όπου προβλέπεται. Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε έγκαιρα για την εξέλιξη στην υπόθεση. Ήδη ο κύριος Έτιγκερ τα συζήτησε σε κάποιες συναντήσεις ε, και κλεισμένων των θυρών. για τη Σλοβακία. Τώρα σας ε, ε, διαβεβαιώ ότι είναι το θέμα το οποίο σοβαρά το εξετάζουμε. Από όταν είχαμε τις ε, πρώτες κατηγορίες, ισχυρισμούς και από τότε που ξεκίνησαν οι συγκεκριμένες διαδικαστικές πράξεις είχαμε επομένως καταγγελίες περί απάτης και ξεκίνησε η Όλαφ τις έρευνες τώρα Όσον αφορά τη διαχείριση, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας τα παρακολουθεί και εποπτεύουμε το πρόγραμμα δράσης και τις πληρωμές. Πάντως έχουμε ελέγχους οι οποίοι είναι εν εξελίξη και οι οικονομικοί κίνδυνοι θα καλυφθούν από την οικονομική δημιουργική παρέμβαση. Βεβαίω και λαμβάνουμε υπόψη το τι γίνεται με το κράτος δικαίου και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Τώρα, όσον αφορά την συνεργασία και τους συνεταιρισμούς θα πρέπει να τα μελετήσουμε για να σας ε, τα πούμε με λεπτομέρειες. Επίσης όσον αφορά την αρπαγή της γης, ε, το ίδιο ισχύει και έχουμε κάποιους ενεργούς ε, γεωργούς που ενέχονται εδώ. Ε, πάντως καταρχήν είναι αυτό εθνική αρμοδιότητα των αρμοδίων κρατικών αρχών. Αυτοί θα πρέπει να καταβάλουν ό,τι πρέπει. Αλλά εμείς παρακολουθούμε προσεκτικά τη λειτουργία του συστήματος. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού ελέγχου είδαμε τι γίνεται με τους φορείς των εκταμιεύσεων των πληρωμών, τι κάνουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές. Και σας τονίζω ότι οι άμεσες πληρωμές καταβάλλονται όχι εις τον κύριο του ακινήτου, αλλά σύμφωνα με τον κανονισμό καταβάλλονται στον χρήστη και ανάλογα με το τι όροι διέπουν την χρήση της γης. αν όλα γίνονται σύμφωνα με τις δέουσες πρακτικές και γίνεται σωστά η διαχείριση. Γιατί έχουμε leasing, χρονομίσθωση για πολλά κίνητα, πολλά κομμάτια γη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εν προκειμένου βρίσκεται να εξελίξει έρευνα στην Σλοβακία. Αν πάντως υπάρχουν ε, άλλες ενδείξεις ότι υπάρχει θέμα και πρόβλημα αρπαγής γης, ε, τότε εάν θεωρηθεί ότι εδώ συντρέχει περίπτωση απάντηση θα ενημερωθεί η Όλαφ και θα ε, επιληφθεί. Αν πάντως είναι θέμα και διαχείρισης και θέμα του ελέγχου, τότε εμείς ασχολούμεθα εμείς κάνουμε τον έλεγχο και έχω να σας πω ότι επίσης βρίσκονται εν εξέλιξη οικονομική έλεγχη στην Σλοβακία αλλά και στη Ρουμανία. Βεβαίω και όταν έχουμε άλλα πιο συγκεκριμένα στοιχεία για αυτές τις διαδικασίες, ε, βεβαίω και θα ενημερώσουμε. και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της έρευνας και αν βεβαίως συντρέχει περίπτωση απάντηση τότε θα είμαστε σε επαφή με την Όλαφ. Μερκοσούρ. Ε, βέβαια. Και υπάρχουν εδώ κάποια στοιχεία στη συμφωνία που αφορούν την προστασία των ευαίσθητων προϊόντων. Και εξασφαλίζουμε ότι οι εισαγωγέ που συμβαδίζουν με τα πρότυπα SPS, ότι λαμβάνεται υπόψη περιβαλλοντική νομοθεσία, ότι αφορά την προστασία του κλίματος. Είναι επίτευγμα αυτή η συμφωνία, γιατί καλύπτει νέα θέματα. Σύστημα ε, αναπτυξιακής ενίσχυσης, ε, λαμβάνεται υπόψη και η Συμφωνία των Παρισίων, καλύπτεται το πρόβλημα της απλής των δασών και υπάρχουν κρατικέ δεσμεύσει για το κλίμα. Παράδειγμα είναι η Βραζιλία. Και σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων έχει δεσμευτεί η Βραζιλία να φτάσει στο 0% τη αποψήλωση των Αμαζόνια. Έχουμε να οξύρωσε 12 εκατομμύρια νεκταρίων Και χρειάζεται να υπάρξει βιώσιμη διαχείριση και να σταματήσει ό,τι αποτελεί παράνομη και μη βιώσιμη πρακτική. Όλα αυτά καλύπτονται από τη συμφωνία. Και βέβαια εμείς θα παρακολουθήσουμε την εφαρμογή της συμφωνίας. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Θα υπάρξουν και άλλες πολλές ερωτήσεις. Είμαι βέβαια κυρία Πένκοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν έχω ρωτήσει. Ευχαριστώ. Ολιβιέ Σαστέλ. Ολιβιέ Σαστέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, εγώ έχω ερωτήσεις, πράγματι. Το 2018 η Κομισιόν ε, επιβεβαίωσε 730 διορθωτικά μέτρα για τη γεωργική πολιτική, 730 πάνω σε 1222 μέτρα που συνολικά είναι οι ενέργειες που προβλέπονται για την ε, μείωση του ποσοστού αυτού και την καλύτερη κατανομή των κονδυλίων, δεδομένων, των επιστροφών στην γεωργική πολιτική και την ε, αγροτική πολιτική. Ποια είναι τα μέτρα για την περαιτέρω απλούστευση της ονομοθεσίας της Ένωσης και τη μείωση των διοικητικών διατυπώσεων για τους αγρότες. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτησή μου. Και επίσης, τα Άγκρι. Τι κάνει με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι μεγάλες ξέρουμε ότι πολλές φορές δεν χρειάζονται βοήθεια. Εν μέρη για τους στόχους ε, απόδοσης και τους ε, δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μείωση μεταξύ άλλων ε, των διαφορών μεταξύ εισοδηματικών ε, μεταξύ του εισοδήματο των γεωργών, για πρόθεση των νεαρών αγροτών κτλ. Και τέλος, οι δείκτες για το ετήσιο ποσοστό χρησιμοποίησης περιβαλλοντικών μεθόδων ε, στις καλλιέργειες. Πολύ αισιόδοξοι οι δείκτες κατά με. Για το 17 και το 18 η Γενική σας Διεύθυνση μιλάει σε μια ανάλυση εξωτερικού εργολάβου που λέω ότι μόνο μικρές ήταν οι αλλαγές στην ε, διαχείριση με εξαίρεση κάποιου συγκεκριμένου τομείς. αυτός ο εξωτερικός ε, μελετητής ποιος ήταν, τι κόστος είχε η μελέτη του και γιατί έγινε η εξωτερική αυτή αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Ίσως ε, να κάνετε εσείς τώρα, κυρία Φανκράμ, την ερώτησή σας. Αν είναι δυνατόν, ναι βεβαίως είναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Ξεκινάω τότε Μπορώ να συμφωνήσω με το τελευταίο σχόλιο του προλαλήσαντα συναδέλφου ό,τι αφορά τη δήλωση και την έκθεση αυτή. Υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις σε ό,τι αφορά ε, ε, τα εισοδήματα των ε, αγροτών πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική όταν μιλάω γιατί σε ό,τι αφορά το στη συνολικό εισόδημα των αγροτών δεν θέλουμε κάποια αύξηση γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πλούσια, πολλές πλούσιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις αλλά θέλουμε να το δούμε ατομικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αγρότης ή η αγρότησα ή συγκεκριμένη μπορεί να είναι φτωχή. Μπορεί το εισόδημα που προέρχεται έρχεται από τη γεωργική παραγωγή να μην είναι τόσο υψηλό. Αλλά πολλέ φορέ οι οικογένειε είναι πολύ εύπορε. Επομένω, πρέπει να τα βλέπουμε καλά τα πράγματα και να τα ξεχωρίζουμε. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά, αν λέω ότι είναι χαμηλά τα εισοδήματα ε, και κάτω από το μισό Αν δει κανεί τι διακοιμάσει, τι παραλλαγέ που υπάρχουν, ότι έχουμε ε, επιχειρήσει εύπορε, πάρα πολύ κερδοφόρε, που είναι πολύ πάνω από το μισό αυτό στατιστικά και οικονομετρικά δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι σωστό και θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να μπούμε σε λεπτομέρειε λεπτομέρειες, να δούμε πόσα άτομα αριθμεί το νοικοκυριό κτλ. κτλ. Και μετά να το σπάσουμε σε ε, κρατήδια ή χώρες κτλ. έπατε επίσης ότι προσπαθείτε και το ρώτησε και ο Βέλγος ε, συνάδελφος ότι προσπαθείτε για τους μικρούς ε, αγρότες να δώσετε ένα μεγαλύτερο μερίδιο επιδοτήσεων, υψηλότερης επιδοτή στήριξη. Σε κάποια κράτη ε, είναι πιο επιτυχής αυτή η προσπάθεια, σε άλλα κράτη όχι. Υπάρχει πλήρης ε, κακό ε, ε, κατάχρηση, μάλλον πολύ κακή κατανομή της, ε, των πληρωμών. Υπάρχουν και μελέτες που το αποδεικνύουν αυτό, το λένε ξεκάθαρα και αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα. Δηλαδή δεν βλέπω να ασχολείστε με την πραγματική αξιολόγηση ε, των ε, επενδύσεων και των επιδοτήσεων μάλλον. Ξέρετε ότι κάποιες χώρες που μπήκαν το 2004 με, τη, με το top-up και τη διαβελιξία μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα ε, επιλέγετε τελικά να εστιάζετε σε λίγες ε, επιχειρήσεις ε, και έχετε άλλους ε, μικρούς εκμεταλλευτές με μισό εκτάριο που τη βγάζουμε 20 ευρώ επιδότηση. Δεν έχει να κάνει αυτό με σωματική υποστήριξη, είναι καταστροφή αυτό και πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Είναι τελείως λάθος η κατανομή των ενισχύσεων. Τελικά τι θέλουμε να πετύχουμε με την γεωρική πολιτική και όλο και μεγαλώνει ψαλίδα. Ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή τα κονδύλια που δίνονται στα κράτη. Τελικά αφήνουμε κάποιους ε, με τα αγορακεπευτικά τους προϊόντα, με τις καλλιέργειές τους να κερδίζουν πολύ περισσότερα από άλλους και τελευταίο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και την προστασία του κλίματος. Ε, αν επιτρέπουμε με τις ενισχύσεις που δίνουμε την ένταση γεωργία στην εντατική καλλιέργεια όταν βλέπουμε ήδη ε, πόσο υψηλέ είναι οι τιμές των αζωτούχων κτλ. Πόσο βιώσιμοι αηφόροι είμαστε ε, περιβαλλοντικά. Ως φορολογούμενοι κάτοικοι ε, των περιοχών αυτών, όταν έχουμε επί δεκαετίες προβλήματα με τη χρήση του νερού, και στο δεύτερο πυλώνα επιλέγει, μάλλον επιτρέπονται κάποια πράγματα. Ξέρω ότι είναι εθνική ευθύνη, αλλά η Κομισιόν και η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Άγκρη θα πρέπει να απαγορεύει αυτά που γίνονται και αυτό θα ήθελα να το ε, κατοχυρώσουμε, να μην επιτρέπουμε στο μέλλον αντίστοιχα φαινόμενα ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, ε, της, ε, του κλίματος. Sorry. Thank you. Uh, I will follow where my colleague uh, basically finished. Uh, the Director General regarding reservations in 2000. Σε σχέση με τις επιφυλάξεις της έκθεσης, οι σχετικές αφορούν για την Τσεχία το τι γίνεται στην κτηνοτροφία, τι γίνεται με κιλομετρίες των ζώων. Πολλές φορές αυτά κυκλοφορούν και δεν είναι βάσιμο. Θα πρέπει να διασταυρώνται αυτές οι πληροφορίες ε, από κράτη, από διάφορους ε, ε, οργανισμούς, γιατί πολλές φορές θα πρέπει να δούμε αν συντρέχει περίπτωση εδώ του να χτυπήσει τον καμπανάκι του κινδύνου. Και έχουμε στον Αντρέι Μπάμπιτ που είναι και πρωθυπουργό και ολιγάρχε. Όμω ε, έχουμε πάρα πολύ σωστή δημοσιογραφία έρευνα εδώ και βέβαια υπάρχουν πολλά κίνητρα για να αναφέρει κανείς τι γίνεται ε, για να μην υπάρχει συγκάλυψη. Νομίζω ότι αυτό είναι μόνο κορυφή του βαγόνου. Κινδυνεύει η ΚΑΠ. Θα ήθελα να μου πείτε Εάν υπάρχει χειραγώγηση από τα κράτη-μέλη όσον αφορά τη διαχείριση, τι ίδιες υπάρχουν ότι για Μάλτα, Ρουμανία, Τσεχία και άλλα κράτη-μέλη, τι γίνεται όσον αφορά την αξιοποίηση, την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τι γίνεται με την σύγκρουση συμφερόντων. Πότε όσα έχετε θα τα δημοσιοποιήσετε όταν στην οριστική τους μορφή. Λοιπόν, κύριε Γενική Διευθυντά, ένα πράγμα θέλω να πω. Ότι εγώ δεν το βρίσκω καλό η Κομισιόν να μας καλεί να καταθέτουμε εμείς συγκεκριμένες περιπτώσεις, ε, να ε, τις γνωστοποιούμε εμείς. Είναι δουλειά της ε, Κομισιόν να ασχολείται με τη Τσεχοσλοβακία. Δεν έχει σχέση με το leasing. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι όλα γίνονται σωστά. Υπάρχουν και διάφορα μοντέλα βέβαια. Αυτό δεν Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να ελέγχετε εσείς πού ακριβώς προκύπτει αυτή η φαρπαγή γης και με ποια μέθοδο. Δεν έχει σχέση με το leasing. Ε, και δεν μπορούμε αυτό να το αγνοούμε. Και ειλικρινά ε, μας το λένε τόσο συχνά τώρα πια οι άνθρωποι, σας το λέω και σκληρά, φοβούνται για τη ζωή τους. Δεν είναι απλά τα πράγματα ε, και η Επιτροπή Κούντ πήγε στην Σλοβακία και στη Ρουμανία και εκεί είναι πάρα πολλέ αυτέ οι περιπτώσεις. Άρα δηλαδή δεν μπορεί κανείς ε, να επαφείται μόνο στι ε, εθνικές αρχές, γιατί ξέρετε κάτι, ε, στα δικαστήρια σε αυτές τις χώρες υπάρχουν πολλές καταγγελίες διαφθορά που συνδέονται με φαρπαγή γη. Ε, κάποια στιγμή πρέπει και η Κομισιόν να πει ότι ξέρει τι γίνεται. Σα το λέω κατηγορηματικά ότι εμεί ω ευρωβουλευτέ δεν μπορούμε να ψάξουμε κάθε μία περίπτωση. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει μια συγκεκριμένη έκθεση από πλευρά Επιτροπή, γιατί όσον αφορά τη διανομή, εκεί υπάρχουν πάρα πολλά κακό κείμενα. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω με το τελευταίο μου σχόλιο, κυρία Πρόεδρε, να σας πω ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς, ε, ότι εμείς περιμένουμε άλλοι να μας τα επισημάνουν. Εμείς ε, βλέπουμε τι γίνεται με τους ελέγχους και οι ε, ελεγκτές μας κάνουν τη δουλειά τους και δεν είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται μόνο στις εθνικές αρχές Υπάρχει κοινή διαχείριση και με τα κράτη-μέλη και οι έλεγχοι γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς λοιπόν κάνουμε τη δουλειά μας, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο ελέγχων για κάθε χρόνο, ελέγχουμε συστηματικά το πώς ε, λειτουργεί το σύστημα. Αν λοιπόν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις από διάφορες πηγές, από τον τύπο, κάποιες επιστολές που στέλνονται σε εμά, ε, γιατί υπάρχουν και γεωργοί που μας στέλνουν επιστολές και ε, λειτουργούμε πάρα αυτά μόλις ε, μας σταλεί, μας επισημανθεί κάποια περίπτωση. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε φήμες, κάποιος είπε κάπου πρέπει να ξέρουμε συγκεκριμένα γεγονότα και μετά και εμείς παρεμβαίνουμε. Εάν λοιπόν υπάρχουν τέτοιου πληροφορίες, με μεγάλη μας χαρά να μας τις δώσετε. Συγγνώμη, λέει πρώτο. εδώ και δύο χρόνια σας ρωτάω για τη Σλοβακία, εντοπίσατε κάτι σχετικό. Σας λέω, στη Σλοβακία κάνουμε έλεγχο. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που ελέγχονται, αλλά δεν μπορούμε να σας τις ανακοινώσουμε τις πληροφορίες, δεν είναι δημοσιοποιήσιμες. Οι έρευνα συνεχίζεται στην Σλοβακία. Στη Ρουμανία προς το παρόν κατά τη διάρκεια των ελέγχων δεν προέκυψε να υπάρχει κάποια περίπτωση υφαρπαγής γης. Και οι γεωργοί δεν διαμαρτυρήθηκαν. Η πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Αλλά σας είπα, πρέπει να έχουμε στοιχεία και μετά θα δραστηριοποιηθούμε. θα συνεχιστεί ο έλεγχος στη Ρουμανία και ε, θα δούμε πώς θα εργαστούμε, αλλά θα εργαστούμε με βάση τους κανόνες. Και αν υπάρχει κάποια απάτη, γιατί αυτό που λέτε ε, είναι παραβίαση κανόνων. Δεν πρόκειται για κοινή γεωργική πολιτική η φαρπαγή γης δεν έχει σχέση με την κυνηγυρική πολιτική. Η πρόεδρος, δεν μπορείτε να δίνετε χρήματα σε κάποιον που έχει αρπάξει γη, να τον χρηματοδοτείτε. εάν είναι παραβίαση κανόνων και είναι ποινική περίπτωση, η Όλαφ πρέπει να το ψάξει, όχι εμείς. Εμείς δεν έχουμε καμία δυνατότητα να παρεμβαίνουμε και αν βεβαίως ε, υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία του συστήματος, εμείς ε, κάνουμε τη δουλειά μας, ε, προσπαθούμε να διασφαλίσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με καθαρές οικονομικές διορθώσεις. Όπως σας είπα, το θέμα αυτό χρήζει περαιτέρω παρακολούθησης και συζητήσεων το προσωπικό μου και εγώ με μεγάλη μας χαρά να συζητήσουμε μαζί σας για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να επανέλθω στα ερωτήματα σχετικά με τον πολύ μεγάλο αριθμό μέτρων ε, που ε, λαμβάνουμε στο πλαίσιο των προγραμμάτων ανάπτυξης. Ε, δεν ξέρω πώς μπορούμε να επιτύχουμε απλούστευση, να βοηθήσουμε τους γεωργούς. Πρώτα απ' όλα προσπαθούμε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, να αλλάξουμε το μοντέλο του πώς λειτουργεί η κοινή ορική πολιτική, να βασιστούμε περισσότερο στην απόδοση, να φύγουμε από την ε, ε, compliance στην απόδοση και αυτό αφορά πολλά μέτρα που εφαρμόζονται. Μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε ε, σε θέματα που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους βασικούς μας στόχους. Βεβαίως όλα αυτά αυτά μπορούν να γίνουν στα πλαίσια της ε, μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται. Όσον αφορά την απλούστευση υπάρχουν ε, πάρα πολλά παραδείγματα, κυρίως ε, στον κανονισμό Omnibus, ο οποίος τώρα εφαρμόζεται παραδείγματο χάρη για τα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν χαμηλό ποσοστό σφάλματος και τα πάνε καλά στους ελέγχους. Εκεί μπορεί να περιστεί ο αριθμός ε, των αγροτών ε, που ελέγχονται από το 3% να πάει στο 1% ή όσον αφορά την χρήση της ε, νέας τεχνολογίας. Αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους, να αντικατασταθούν οι επιτόπιοι έλεγχοι με ελέγχους εξ και αυτό σίγουρα θα διευκολύνει τη ζωή των γεωργών. Όσον αφορά τώρα το θέμα που έχει σχέση με τις διαφορές που διαπιστώνονται στο εισόδημα ανάμεσα στους μικρούς και τους μεγάλους γεωργούς. οι πληρωμές ε, στους γεωργούς γίνεται με βάση την έκταση της ε, γης. Βεβαίω, οι μεγαλύτερε εκτάσει χρηματοδοτούνται περισσότερο. Παίζει ρόλο και το θέμα του κλίματος. Είναι σημαντικό να καλλιεργείται κάθε εκτάριο. Ε, καταμπάλλονται πολλές προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιωθεί η κατανομή των άμεσων πληρωμών. Για πολλά χρόνια προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε το κάπινγκ, την, τη μέγιστη ε, χρηματοδότηση ανακαλλιέργεια, ανα εκμετάλλευση μάλλον, και πάλι τώρα λέμε μέγιστη πληρωμή ανα αγροτική εκμετάλλευση να πούμε 100.000 ανώτατο όριο αναγεωργική εκμετάλλευση. Αλλά για να περάσει αυτό σε Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πρέπει να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περιμένουμε λοιπόν την υποστήριξη και των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει μια πολιτική που προβλέπεται, και για το μέλλον η δυνατότητα να υπάρχει υψηλότερη χρηματοδότηση για τα πρώτα εκτάρια ε, σε κάποια κράτη λειτουργεί αυτό, αλλά πάλι οι κράτη ζητούν ε, το, το κάπινγκ, το, το ανώτατο όριο. Εμείς θέλουμε να υπάρχει καλύτερη διανομή. Πράγματι, έχετε δίκιο, στατιστικά και με τις έρευνες, τις στατιστικές, ε, ε, τα στοιχεία μπορούν να ερμηνευτούν και διαφορετικά. Αλλά θα ήθελα να σας πω, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αν πάρουμε γενικότερα τα στατιστικά δεδομένα ε, η χρηματοδότηση ανά εκτάριο για τις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις μειώνεται όσο μεγαλώνει ε, η γεωργική εκμετάλλευση. Τα πρώτα εκτάρια χρηματοδοτούνται περισσότερο από ότι τα τελευταία. Αυτό φαίνεται και στην ε, έκθεση ετήσιας ε, την ετήσια έκθεση. Ίσως το χάσμα να μην μειώνεται αρκετά γρήγορα, αλλά το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις πληρωμές που αφορούν κράτη-μέλη με πολύ ψηλή χρηματοδότηση ανά εκτάριο, όπως είναι η Σλοβακία, το χάσμα ανάμεσα στις διάφορες χώρες μειώνεται. Μήπως μπορώ να σας ζητήσω σιγά-σιγά να ολοκληρώσετε. Θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στις ε, περιβαλλοντικές φιλοδοξίες. Είπατε ότι η έκθεση είναι υπερβολικά αισιόδοξη. Νομίζω ότι εστιάζουμε στις ε, πληροφορίες που έχουμε ένα σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου που συγκεντρώνει στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Και θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που λειτουργούν αρκετά καλά. Ε, Παραδείγματο χάνει το 30% ε, του αγροτικού δυναμισμού είναι υπό το καθεστώ permanent patcher, των ε, μόνιμων ε, ε, βοσκοτόπων. Και κατά τα άλλα, η πολιτική που εφαρμόζουμε περιλαμβάνει κάποια στοιχεία πρασινίσματος. Πρόσφατα αποφασίστηκε να μην χρησιμοποιούνται ζυζανιοκτώνα σε παραγωγικές εκτάσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική, αλλά για το μέλλον ε, παραμένουν πολλές προκλήσεις και γι' αυτό εμείς προτείνουμε να εμβαθύνουμε και να εστιάσουμε στα αποτελέσματα, όχι στη συμμόρφωση αλλά στα αποτελέσματα. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω βέβαια πάρα πολλά να πω και για την οριζόντια ερώτηση που ετέθη ε, σχετικά με τη δήλωση για την ποιότητα της αναφερόμενης απόδοσης. Θέλω να σας πω ότι η δήλωση στην ετήσια έκθεση είναι απόλυτα σαφής. Εγώ αναλαμβάνω της ευθύνης μου για το θέμα της απόδοσης. Ένα μεγάλο κομμάτι της αφορά την απόδοση και στην ε, έκθεσή μας αναφερόμαστε σε βασικούς δείκτες απόδοσης, αλλά βέβαια όσον αφορά τα άλλα θέματα, θα ήθελα να σταματήσω και να ε, επανέλθω αυτά που είπε ο κύριος Πάκα πριν από μένα. Είμαι σίγουρη ότι για τη Γεωργία υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μας απασχολούν ακόμα. Νομίζω θα επανέλθουμε έτσι. Αυτή την εντύπωση έχω. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το γύρο, τον πρώτο γύρο και θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες. Πάμε στον επόμενο ομιλητή. Κύριος Μάκλεμερ, παρακαλώ μην ξεπεράσετε τα πέντε λεπτά αν μπορείτε, γιατί αλλιώς θα καθυστερήσουμε ακόμη περισσότερο. Vorsitzende, guten Morgen. Ähm, äh, herzlichen Dank meinerseits auch. Ich werde mein Bestes tun. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υπάρχει χώρος και για ερωτήσεις. Αξιότιμοι βουλευτές. Αγαπητοί βουλευτές της Επιτροπής Κοντ, θα εστιαστώ εις δύο θέματα. της επιδόσης, απόδοση μας και από την άλλη μεριά στις εγγύησεις. Ε, τώρα, όσον αφορά τις επιδόσεις μας από πλευράς χρηματοοικονομικής για τα δύο ταμεία αρμοδιότητός μας, η RDF και Ταμείο Συνοχής, δηλαδή Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ταμείο Συνοχής, έχουμε τώρα ε, δύο την να σας ε, αναφέρουμε το θετικό είναι ότι μέχρι τώρα έχουμε ένα ποσοστό επιλογής για συγκεκριμένα προγράμματα αυτών των δύο ταμείων είναι πάνω από 80% των υπαρχόντων μέσων και πόρων. Όμως, λιγότερο θετικό είναι το άλλο νέο, δηλαδή το τι γίνεται όσον αφορά το ποσοστό εκτέλεσης και υλοποίησης της πολιτικής. Αυτό είναι μετρήσιμο ε, με τις ε, τελικές καταβολές προς τα κρατημέλη. Εδώ είμαστε σε ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο. Είμαστε λίγο πιο κάτω από το 1 τέταρτον του υπάρχοντος ποσού, παρά το ότι πλησιάζουμε στο τέλος της εξαετίας αυτού του πλαισίου, του δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό είναι ελάχιστα ικανοποιητικό και σας επισύρω την προσοχή στο εξής. Πρώτον, η πρώτη διάσταση του φαινομένου. Έτσι, έχουμε σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την χρηματοοικονομική διαχείριση σε επίπεδο υπολογισμού της Ένωσης. Και τώρα είναι αναπόφευκτο ότι πάνω από 50% των ε, κονδυλίων πολιτική θα πρέπει να καταβληθούν στην επόμενη χρήση. Άνω του 50%. Δεύτερον, και κατά γνώμη μου αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν προκύπτουν τα ωφέλη που προσδοκούν οι πολίτες από την πολιτική συνοχή. Μερικά παραδείγματα. Γι' αυτό σας λέω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ως μέτρο απαραίτητο προοδευτικά να επιστρέψουμε σε περισσότερη δημισιονομική, χρηματοοικονομική πειθαρχία. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία κύριε. Και συγκεκριμένα να επιστρέψουμε στο N+. Αυτός ο κανόν που ίσχυε στο παρελθόν τώρα. Γιατί αναφέρομαι στους πολίτες, αν δούμε συγκεκριμένα ποιοι είναι οι δείκτες των επιδόσεων, πού βρισκόμαστε σήμερα δημιουργία απασχόληση σε σχέση με τι ΜΜΕ. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον κόσμο, ακριβώ πόσε θέσει εργασία ε, ενθαρρύνουμε να δημιουργηθούν. Ε, στο τέλο του 2018 ήμασταν στι 43.000 θέσει απασχόληση. Τώρα ποια είναι η προσδοκία για το σύνολο τη περίοδου. Και εδώ πέρα είμαι πάρα πολύ συντηρητικό στα όσα λέω. Μιλάμε για 500.000 θέσει εργασία, επομένω, δεν έχουμε φτάσει ούτε το 1 δέκατο ω αποτέλεσμα σε σχέση με τι συνολικές προσδοκίες. Δεύτερο παράδειγμα, τα ερευνητικά προγράμματα μεταξύ επιχειρήματος και ερευνητικών ιδρυμάτων. Περίπου 6.000 τέτοια προγράμματα έχουμε, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί για το σύνολο της περίοδου. Ο στόχος ήταν πάνω από 60.000 προγράμματα. Και εδώ πάμε στο ότι βρισκόμαστε στο 1% του προσδοκομένου και θα μπορούσα να συνεχίσω με αυτό αυτό πνεύμα. Αλλά φαντάζομαι ότι κατέστην σαφή. Τώρα να σας επίσης την προσοχή σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Από τι σημαίνει εξέλιξη ότι δηλαδή έχουμε ένα πλαίσιο για την επίδοσή μας που είναι στεγανό. Δεν βγάλαμε αυτά από το κεφάλι μας, δεν, δεν είμαστε θροβάμενες έχουμε αυτό το στεγανό πλαίσιο και επίσης ε, το σύστημα υποβολής εκθέσεων των κρατών μελών και διαβεβαιώ τον κύριο Σαστέλ ότι η αξιοπιστία των δεδομένων των επιδόσεων από όλες τις διαχειριστικές αρχές είναι κάτι το οποίο περνάει από ελέγχους σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο κομισιών. Και όποτε υπάρχουν προβλήματα, τότε μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και την αναστολή των καταβολών μέχρι ότου η αξιοπιστία αποκατασταθεί. Και υπάρχουν τέτοιε περιπτώσει σήμερα. Να έχουμε αναστείλει πληρωμέ εξ αυτού του λόγου. Ότι δηλαδή τα στοιχεία για τι επιδόσει δεν ήταν αξιόπιστα ή δεν είναι αξιόπιστα. Για να δούμε τώρα ε, τι έγινε, ε, τι έγινε στο τελευταίο δίμηνο ας πούμε, για να μπορεί να δείτε τι γίνεται με αυτό το 6% ως αποθεματικό και να δούμε τι έγινε όσον αφορά την αναδιανομή των ε, πόρων ε, γιατί σε μερικού τομείς έχουμε ιστερούσα επίδοση. Δεν θα μπω τώρα στα διαδικαστικά των ε, εγγύσεων 14 έως 2020. Γίνανε πολλές αλλαγές σχετικά το παρελθόν για να δούμε τι λάβαμε υπόψη ούτως ώστε να θωρακίσουμε αυτό το σύστημα ιδίως τους τίσους λογαριασμούς που μας διαβιβάζουν και που καλύπτουμε 2016 και 2017. Είχαμε 175 τίσιους λογαριασμούς να ελέγξουμε σε σχέση με 35 την προηγούμενη χρήση. Και αυτό σας δείχνει πόσο αργά ξεκίνησε η διαδρομή, η πορεία αυτή. Και με βάση αυτά, τσεκάραμε αυτούς 185 λογαριασμούς και επί τη βάση εξολόγηση του κινδύνου είδαμε τι γίνεται στα κρατημέλη για τις επιδόσεις όσον αφορά το 1 τέταρτον αυτών των ε, επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οπότε είπαμε ότι στην ετήσια έκθεση έχουμε βάλει το τι γίνεται με τον κίνδυνο και τις πληρωμές. Κάτι λιγότερο από 2%. Και όταν υπογράψαμε την ετήσια έκθεση του ελέγχου, ακόμα υπήρχαν κάποιες ε, περιπτώσεις κάποιων επιληψίμων περιπτώσεων όσον αφορά την αξιολόγηση. Και στο χειρότερο σενάριο ο κίνδυνος θα ανέβαινε στο 2,7% σε κάθε περίπτωση. Οπότε καταλήξαμε ότι ο κίνδυνος για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πάνω από το 2% τότε ζητήθηκαν επιπλέον διορθώσεις. Αυτό έγινε σε 29 προγράμματα. Τώρα τα είδη των σφαλμάτων. Έχουμε καλύτερη ενημέρωση οπότε στο παρελθόν γιατί έχουμε μια πια παγιωμένη τυπολογία συνήθως το σφάλμα αφορά μη επιλέξιμη δαπάνη 40% των σφαλμάτων σχετίζεται με τέτοιες μη επιλέξιμες δαπάνες τώρα δεύτερη ομάδα σφαλμάτων αφορά λάθη στους κρατικούς διαγωνισμούς Συνήθω αυτό είναι διαδικαστικά λάθη κατά το εντρίδων των περιπτώσεων. Αυτά είναι τα κυρία λάθη τώρα. Έχουμε δύο επιφυλάξει για την περίοδο 2014-2020 όσον αφορά 30 προγράμματα. Δηλαδή το 1 τέταρτο του συνόλου των ε, προγραμμάτων και επίσης για το 2007 έχουμε 13 για 80 προγράμματα αλλά και είπαμε είναι άλλη διαδικασία και η τελική καταβολή γίνεται όταν ε, έχουμε εξασφαλίσει ότι έχει πέσει το ποστό σφάλματος κάτω από το 2%. Επομένω δεν πρόκειται περί χρηματοοικονομικής ε, επιφύλαξης εν προκειμένου. Ό,τι άλλο θέλετε, θα σας τα πω στις ερωταπαντήσεις. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω γρήγορα να κάνω τις ερωτήσεις μου και να κάνω και ένα είδος ε, συνόψησης ε, σε ό,τι αφορά το ελεγκτικό καταλήγει σε περιθώριο όντως πάνω του 5% και κάτω το 2% λέει η Κομισιόν. Υπάρχει μία αντίφαση εδώ, δεν καταλαβαίνω που οφείλεται. Σε, που, σε τι οφείλονται οι διαφορές ε, ε στις υπολογισμούς μεταξύ ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ και Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ποσοστό σφάλματο. Και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα που είναι σημαντικό ποσοστό ε, πρόβλημα και πού είναι ε, τα προβλήματα με τα χρηματοδοτικά μέσα, θα ήθελα να μου πείτε. Και για το 2018, 258 προγράμματα και 10 με την έμπλωση ε, καθήλυνα αρμόδιο έχουν υποβάλει λογαριασμούς μπλα μπλα μπλα μέχρι την 1η Μαρτίου. Δέχτηκε 242 επιστοποιημένους λογαριασμούς. Αλλά δεν μπορείτε να πείτε τίποτα για τα πακέτα διασφάλισης ε, μέχρι το 18 γιατί συνεχίζετε τις επαληθεύσεις. ΣΝΔ um, First, uh, Πένκοβα, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λεμέτρα, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Αρχίσατε με ένα σημαντικό Ε, χαμηλά ποσοστά απορρόφησης για το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Δώσατε επικαιροποιημένα στοιχεία. Το ερώτημά μου είναι, παίρνετε όμως συγκεκριμένα μέτρα. για να λυθεί το πρόβλημα της απορρόφησης από τα κράτη-μέλη, ώστε να μπορούν να ωφελούνται με κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επενδύσεις και αν υπάρξει κάποια καθυστέρηση. Υπάρχει κάποιο ειδικό μέτρο ή μπορείτε να βοηθήσετε με κάποιο τρόπο να χρησιμοποιούνται με τον πλέον αποδοτικό τρόπο τα κονδύλια. Και το δεύτερο αφορά τον κύριο Λεμέτρα αλλά και τον επόμενο, τον κύριο Κόρτε. Σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου του Μαΐου, 72% της απάτης λέει προέρχεται από τα διαθετικά επενδυτικά ταμεία. Τι μέτρα λαμβάνετε για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Και για τον κύριο Κόρτε βέβαια πιο πολύ είναι το ερώτημα αυτό. Υπάρχει λόγος για την αναβολή της κοινή ε, στρατηγικής καταπλήμψης απά της Ολιβιέ Σαστέλ. Ε, Madame la Présidente, deux questions, partiellement. Εν μέρει το ακούσει σε ό,τι αφορά την, ε, δυνατότητα, την ε, ικανότητα απόρρωση που δεν είναι η βέλτιστη. Τεχνική βοήθεια για ε, κράτη-μέλη. Πρέπει να βελτιωθεί, να χρηματοδοτηθεί καλύτερα. Ο προπολισμό τη Ένωση πρέπει να προβλέψει επιπλέον κονδύλια για την καλύτερη κατάρτιση αυτών σε χώρες που έχουμε προβλήματα για να υπάρχει καλύτερη δυνατότητα απορρόφησης. Δεύτερη ερώτηση. Κυρία Πρόεδρε, το ξανά πάμε και αυτό. Ε, το είπατε και εσείς, χρηματοδοτικά μέσα. Σήμερα βλέπουμε σημαντική διακύμανση ανάλογα με τα κράτη-μέλη. Κάποιες φορές 10-12% ε, διαφορά, κάποια δεν έχουν καν χρηματοδοτικά μέσα. Τι εκτιμάτε εσείς. Ιδίω από τη στιγμή που έχουμε και σημαντικά σφάλματα στα χρηματοδοτικά αυτά μέσα. Και πώς διορθώνονται να μου πείτε. Ευχαριστώ. Und Viola von Kramon zum Abschluss. Thanks a lot for your report. Κυρία von Kramon, για να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ την εκθεσή σας. Παρόμοια γραμμή και ειδική μα ερωτήσει όπω οι σοσιαλιστέ και το Ρινιού. Χαμηλά ποσοστά απορρόφηση πρώτα. Φυσικά μα ανησυχεί όλου αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να υπηρετούμε του πολίτε. Το είπατε κι εσεί. Πώ θα του υπηρετούμε όμω, αν δεν μπορούμε να αγγιθούμε την απορρόφηση των κονδυλίων. Υπάρχουν νέες μετρήσεις, ιδέες για να χαμηλώσει, μάλλον να υψηλώσει, η, να βελτιωθεί η απορρόφηση. Ε, backlog, I would like to Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την ε, εκτέλεση των ε, τιμολογίων, την πληρωμή, θα δοθεί κάποιο, θα δοθούν κονδύλια από εσά, έχετε προβλέψει κάτι εσείς, η Κομισιόν εν γέννη, όταν έρθουν τα εντάλματα και για τα διαφορετικά αυτά ποσοστά σφάλματος. Το να χρησιμοποιείτε το residual risk ε, ε, και να έχετε άλλα στοιχεία από την Κομισιόν. Είναι ένα πρόβλημα. Σχεδόν 13 διαφορετικά ποσοστά βλέπουμε. Αυτό δεν βοηθά να υπάρξει σαφήνεια, άρα ε, αυξάνει τη σύγχυση σε ό,τι αφορά και τη διασφάλιση. η έκθεση απαλλαγή λέει ξεκάθαρο του Κομισιόν. Πρέπει να πάψει να χρησιμοποιεί διαφορετικά ε, ποσοστά σαν από αυτά που χρησιμοποιεί το ελληνικτικό. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι και διαφανεί σε σχέση με το τι κάνει, το τι πληρώνει ο ευρωπαϊκό Υπολογισμό, τώρα είναι η ώρα. Τι έχει κάνει η Κομισιόν και τι μπορείτε να κάνετε εσεί στο πλαίσιο τη εντολή σα και αν δεν έχετε κάνει κάτι, γιατί. Ευχαριστώ για την ερωτή σα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τους ε, υπόλοιπους ε, βουλευτές. Ε, θα προσπαθήσω γρήγορα, γρήγορα να απαντήσω. Θα σχολιάσω αυτό που είπατε για το ελεγκτικό συνέδριο και το ποσοστό σφάλματος. Όταν δημοσιοποιηθεί θα σας δούμε, θα σας εξηγήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Θα θέλουμε να δούμε όπως πρώτα την έκθεση του ελεγκτικού για να δούμε γιατί υπάρχει αυτό το διαφορετικό ποσοστό. Uh, the percentages I have been mentioning today. Uh... Αν υπάρχει διαφορά από τα ποσοστά που σας ανέφερα, που δεν θα αλλάξουν, και τα ποσοστά του ελεγκτικού που όπως έλεγα στην έκθεσή του που θα ε, δημοσιοποιήσει λίγο το ελεγκτικό συνέδριο αν υπάρχουν διαφορές θα προσπαθήσουμε να σας εξηγήσουμε. Τώρα τα προγράμματα, τα προβλήματα μάλλον που εντοπίζονται στα χρηματοδοτικά μέσα. Δύο ειδών κυρίως είναι. Το πρώτο έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση, πώς λειτουργεί τι γίνεται με τις προστοβαρείς πληρωμές μας. Προκαταβολές, αν θέλετε, στα χρηματοδοτικά μέσα. Και τι γίνεται από τις διαχειριστικές αρχές. Τι τα κάνουν αυτά τα χρήματα. Τα στέλνουν αμέσως ή αργότερα στους ε, φορείς που διαχειρίζονται αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα. Μάλλον δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό. Τελικά, ένα θέμα χρόνου, λίγων μηνών και μετά λύνεται το πρόβλημα. Και για μια συγκεκριμένη περίπτωση πέρυσι γνωρίζουμε ότι υπήρξε αυτό το πρόβλημα. Όμως η βασική πηγή σφαλμάτων πιο σοβαρή και έχει να κάνει με το τύπο της επιχείρησης που στηρίζεται από εγγύηση και δάνη. Παραδείγματο χάρη, να δούμε τι γίνεται με τις ΜΜΕ και τα σχετικά κριτήρια. Υπήρξαν κάποιες διαφωνίες κατά το παρελθόν μεταξύ ημών και του ελεγκτικού συνεδρίου, διαφορές ως προς την ερμηνεία. Γιατί λέει ορισμό ότι περισσότερο υποστήριξη, the majority, η περισσότερη υποστήριξη, πρέπει να πηγαίνει στις ΜΜΕ. Αυτό αφήνει όμως περιθώρια ερμηνείας. Αυτή η πλειοψηφία, αυτή το μεγαλύτερο μέρος, τι αφορά, εγγυήσεις, δάνεια, τι αφορά αυτό το majority. Και έχω να αναφέρω θετικές εξελίξεις Ιδίω ό,τι αφορά την πρόσβαση στι πληροφορίε που χρειαζόμαστε, αλλά και εμεί και το ελεγκτικό βέβαια. ώστε να γίνονται σεβαστοί από αυτά τα μέσα όλοι οι κανόνε. Και οι διχειριστικέ αρχέ επίση θέλουμε να σέβονται όλε τι ε, όλους τους κανόνες ε, για το όταν ε, δίνουν τα χρήματα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. υπάρχουν υποσπαθητικές εξελίξεις, αλλά για να μην ειλικρινής, Δεν νομίζω ότι προκύπτει από όλα αυτά ότι υπάρχει κάποια ε, δομική αδυναμία στα χρηματοδοτικά μέσα ή δεν ε, δεχετεύονται σωστά τα κονδύλια, άρα δεν θα έπρεπε ίσως να δίνονται σε χρηματοπιστωτικά μετά. να δίνονται αλλού. Ε, επομένως, νομίζω ότι χρηματοδοτικά μέσα και σήμερα και στο μέλλον είναι σημαντικά. Είναι το 11% των ποσοστών σφαλμάτων και είναι πάνω από το 11% των πληρωμών σίγουρα που κάνουμε. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι δυσανάλογο. Ε, ε, on, um, the 2017... Για τους οργανισμούς 17-18. Δεν έχει τελειώσει δουλειά μας. Καλά τα είπατε, κυρία Πρόεδρε. Κάναμε την ε, επανεξέταση, την ανάλυση όλων των λογαριασμών που έχουμε λάβει, αλλά εξακολουθεί ε, να χρειάζεται και επιτόπου έρευνα. Εμείς δεν είμαστε ε, αυτοί που κάνουμε το έργο των ελεγκτών, ε, των διαχειριστικών αρχών, δεν έχουμε τελική εικόνα για την εκτέλεση των λογαριασμών 17-18 ακόμα. Κυρία Πένκοβα. Εστιάσατε αρχικά στην απορρόφηση και ρωτήσατε τι κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις δυνατότητες απορρόφησης. Ακούστε, στην τρέχουσα περίοδο πράγματι θέσαμε σε ισχύ σημαντικά μέσα στήριξης. Το πρώτο, που είναι και από το 2014, είναι το λεγόμενο πλαίσιο ευθυνών αρμοδιότητων. Τι περιλαμβάνει αυτό, περιλαμβάνει τις αρμοδιότητες και τις δεξιότητες που θα έπρεπε να έχουν τα μεμονωμένα μέλη των διαχειριστικών αρχών ή των ε, ελεγκτικών αρχών. Ένα είδος πίνακα με το τι θα έπρεπε να... Ποια θα έπρεπε να πληρούν όλοι αυτοί που εργάζονται στις διαχειριστικές αρχές και ανατοπίζουν ε, τυχόν αδυναμίες. Και αν υπάρξει πρόβλημα με τις δεξιότητες θα πρέπει να μπορούν να τις εντοπίζουν και να τις διορθώνουν οι υπεύθυνοι. Τεχνική βοήθεια ρώτησε ο κ. Σαστέλ. Υπάρχει αυτό στα κράτη-μέλη. Για τη χρηματοδότηση των διαχειριστικών συστημάτων. 40% μάλιστα επί του συνόλου του προπολογισμού. Άρα μιλάμε για μεγάλα ποσά. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξοπλίσουν τα χρήματα αυτά. Για να υπάρξει βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Προσπαθούμε ακόμα όμως να παρέχουμε και άμεση βοήθεια, πέραν της τεχνικής βοήθειας. Υπάρχει κεντρικό προπολογισμό παροχή βοήθεια και από αυτόν χρηματοδοτούμε τη υποστήριξη από ε, εγνωσμένου κύρους, ειδικού κτλ. Και αυτοί πηγαίνουν και εκπαιδεύουν επιτόπου. Ε, ένα παράδειγμα σας λέω, υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει και ελέφαντας στο δωμάτιο, που είναι το Jaspers. Χρηματοδοτούμε στο ύψος των 32 εκατομμύριων το χρόνο. Yeah, especially major projects. And they can turn to this uh, service free of... Και είναι και ελεύθερη, είναι δωρεάν η χρήση της υπηρεσίας. Αρκεί να λάβουν πρωτοβουλία. Άρα υπάρχουν πολλά που γίνονται. Το ότι υπάρχει λοιπόν ε, χαμηλό ποσοστό απορρόφησης οφείλεται στο ότι είναι πολύ χαλαροί οι κανόνες. Όχι ότι είναι γενός ε, ελαττωματικό το σύστημα. Ε, αυτό θέλω να το καταρρύψω ως επιχείρημα. Πρέπει να εφαρμόζονται καλύτερα οι κανόνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την απάτη. Και να αναφερθώ και σε μια πρόσφατη έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου που ε, μελετά το τι έγινε στην τρέχουσα περίοδο. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Τα κράτη-μέλη τήρησαν τους ενισχυμένους κανόνες ώστε οι μηχανισμοί εντοπισμού απάτης να ενσωματωθούν στα διάφορα διαχειριστικά βήματα και διαδικασίες. Και επίσης το βλέπουμε και στο πλαίσιο των ε, συστημικών ελέγχων στα κράτη-μέλη. Είναι καλή προσέγγιση των κρατών μελών για την πρόληψη και αποφυγή απάτης και έχουμε δώσει καθοδήγηση βέβαια και στα κράτη-μέλη στην αρχή της περίοδου επ' αυτού. Βέβαια, αναγνωρίζουμε ότι είναι ένας κινούμενος στόχος αν αλλάζουν οι κανόνες και έχουν αλλάξει κανόνες στον ταυτιστικό συμφερόντων. Άλλαξαν πέρυσι τον Αύγουστο. Και είναι μια κατηγορία στο πλαίσιο της απάτης εν γέννη. Τα κράτη-μέλη από τον Οκτώβρη Έχουμε αρχίσει επαφές και ήδη έχουμε κάνει πολλές, έχουμε διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις και για να γίνει πιο σαφής ορισμός και για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματα διαχείρισης στην αλλαγή. Βέβαια, φυσικά δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη. Παρακαλώ, μήπως μπορείτε να ολοκληρώνετε. Ναι, ναι, βεβαίως, με συγχωρείτε. Ναι, μάλλον μακρηγορώ. Πλατιάζω. Πώς θα βελτιώσουμε στο μέλλον την απορρόφηση. Αν διακτηνιστώ στην επόμενη ε, περίοδο προγραμματισμού ε, πιστεύω θα υπάρξει ένα άλμα για την απορρόφηση. Δηλαδή τι είναι απαραίτητο εδώ. Έχουμε τον ΙΣΙΝ 2 νομίζω ε, ως στόχο γιατί αλλιώς θα είμαστε πολύ αργοί. Και έχουμε προτείνει κάποια μέτρα πλούστευσης που καθιστούν πολύ εύκολη την επιτάχυνση τη κατάσταση. Το πρώτο μέτρο, δεν αλλάζουμε τα συστήματα. Χρησιμοποιούμε και για την προσεχή περίοδο τα σημερινά. Ο εμπροστοβαρής επενδύσει δεν γίνονται κτλ. Το δεύτερο μέτρο θέλω να τονίσω είναι ότι ξε... μάλλον διευκολύναμε τη συνέχιση των προγραμμάτων που έχουν ξεκινήσει αυτή την περίοδο να συνεχιστούν και στην επόμενη. Για να μην ξεκινάμε από το μηδέν. Σχέδιο χρηματοδότησης της καθυστέρησης. Μετά το 20 θα έχουμε πολλά προγράμματα. Ήδη λέγεται πολλά στο, στην πρόταση για το πολιετές. Η πρόταση για το πολιετές που κάναμε περιλαμβάνει οροφές πληροφών για το 2021 2021-2023 που είμαστε σίγουροι έτσι θα μπορούν τα κράτη-μέλη να πληρώνουν εγκαίρω. Και σε ό,τι αφορά τον εξορθολογισμό ποσοστών σφαλμάτων, νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Είπατε 13 διαφορετικά ποσοστά. Αυτό ήταν για πέρυσι. Φέτο έχουμε πολύ λιγότερα. Όμω, αν μπορούμε ακόμα να τα περιορίσουμε, να μην το μελετήσουμε. Βεβαίω και θα το κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και για τις διεξοδικότατες αυτές απαντήσεις αλλά πρέπει να προχωρήσουμε στον επόμενο, στον επόμενο Γενικό Διευθυντή, ο του Κόρτε. Αλλά σας, πρέπει να σας περιορίσω λίγο, διότι δεν θα μπορεί να ρίξει καν το στόμα το τελευταίος Γενικός Διευθυντής ε, πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη συνέντευξη. Παρακαλώ, λοιπόν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Νομίζω ότι μπορώ να είμαι σύντομο, γιατί ο αγαπητός συνάδελφος Μάρκ είπε πολλά από αυτά ε, τα οποία θα να πω και τα οποία αφορούν και το δικό μου τομέα. Ω ΓΑΜΑ Απασχόληση είμαστε πλήρω ενταγμένοι στην ε, πολιτική συνοχή και έχουμε κοινού μηχανισμού με του συναδέλφου τη DG ε, Περιφερειακή Πολιτική τη Γενική Διεύθυνση τέλο Και. Αν θέλουμε να βρούμε την οριοθέτηση, θα μπορούσαν να πει κανεί ότι η διάκριση γίνεται ότι εμείς επενδύουμε στον άνθρωπο και ήταν πολλά τα επιτεύγματα χάρη στις επενδύσεις του κοινωνικού ταμείου ε, όσο κράτησε η κρίση και έχω και κάποια θεμετικά στοιχεία να σας πω και επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια πρόταση φιλόδοξη για το επόμενο δημοσιακό πλαίσιο για το κοινωνικό ταμείο ΣΥΝ όπως το ονομάζεται από τα δισεκατομμύρια σε 101. Έχουμε 215 προγράμματα που τρέχουν τώρα με το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο για τους μη προνομιούχους. Επίσης ε, ασχολούμαστε και με τη συνεργασία με το Ταμείο Προσαρμογής στην Προνομιοποίηση. Τώρα να σας πω τι γίνεται για αγγίσεις και επιδόσεις τώρα στον αφορά τις εγγύησεις όπως γνωρίζετε καλά χάρη στις βελτιώσεις του νομοθετικού πλαισίου για την περίοδο 14 έως 20 το μοντέλο μας τώρα κίστηκε σημαντικά. Τελικά πάντως και τα ακούσατε από τους συναδέλφους και θα το ξαναακούσετε τα κράτη-μέλη τελικά έχουν την ευθύνη της υλοποίησης. Όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έχουμε αυτόν τον κανόνα του 10% της ε, ε, κράτησης για τους ετήσιους ε, διακοπή, αναστολή και επίσης για το κοινωνικό ταμείο έχουμε την ευξημένη χρήση των επιλογών ε, απλούστευσης. Και όλα αυτά τώρα ξαναείπαμε τα συστήματα της διαδικασίας μας. Οπότε έτσι εξασφαλίζεται ότι γίνεται η ορθή χρήση των κονδυλίων και σύμφωνα με τους στόχους που εσείς έχετε θέσει και όπως θα δείτε και από την εκθεσή μου είμαι πεπισμένος ότι λειτουργεί καλά το καινούργιο σύστημα ωφελεί όλο ένα περισσότερο όσον αφορά την ε, το θέμα της εγγύησης. Ε, βέβαια, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων, αυτό και σας ενδιαφέρει. Ε, όχι, δεν είναι όλα καλά. Υπάρχει αυτό το περιθώριο βελτιώσεων. Μην επαναλάβω όσα είπε ο κύριος Λεμέτρα, γιατί έχουμε παρόμοια θέματα. Βέβαια, ισχύει ότι τελικά το μοντέλο μας εδράζεται στο τι κάνουν οι εθνικές ελεγκτικές αρχές. Και γι' αυτό και η Γενική Διεύθυνση έχει επιφύλαξη 28 επιφυλάξεις για 205 προγράμματα. Κοινωνικό Ταμείο, πρωτοβουλία για απασχολήση των νέων και τρεις όσον αφορά το Ταμείο για τους ε, μη προνομιούχους. Ε, Είπαμε ότι υπάρχουν ε, κάποια θέματα σε κάποια σημαντικά ζητήματα και μπορείτε να, το δείτε με δύο τρόπους. Είπαμε 28 επιφυλάξεις για 215 προγράμματα. Ε, δεν είναι και λίγο όλο αυτό. Επίσης σας δείχνει ότι το σύστημα λειτουργεί. Εφαρμόζουμε αυστηρά τους κανόνες, αποπτεύουμε ε, και γι' αυτό εναντί της αρχής του προπολογισμού έχουμε τις απαραίτητες εγγύσεις και θέλουμε βέβαια να εξεταστεί γιατί υπάρχουν επιφυλάξεις και πώς τα κράτη θα λύσουν τα προβλήματα που οδήγησαν σε αυτές τις επιφυλάξεις. Τρία την έχω να σας αναφέρω. Έχουμε ακόμα πάρα πολλές επιφυλάξεις. Πρώτα-πρώτα έχουμε κάποια προβλήματα που σχετίζονται με τα συστήματα επαλήθευσης της διαχείρισης προβλήματα με τους δημόσιους ε, διαγωνισμούς, λιγότερο όσον αφορά το περιφερειακό ταμείο και κάτι άλλο το οποίο ανακαλύφθηκε φέτος. Τους ελέγχους επιλεξιμότητας αυτών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για απασχόληση των νέων. Είναι και θέμα του timing. Ενοχλητικό, δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε τίποτα. Κάποιες ειδικές αρχές δεν ολοκλήρωσαν τον έλεγχο εγκαίρως για να μπουν αυτοί στους ετήσιους ε, λογαριασμούς. Ε, αυτά μας ε, προβληματίζουν, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και όλα αυτά τα λάβουμε υπόψη, υπόψη για το μέλλον. Σας λέω ευθύς αμέσως ότι όταν υπέγραψα την έκθεση από τις 28 επιφυλάξεις έχουν ήραμε, έχουμε τέλο πάντων άρει μέχρι τώρα τι 7 επιφυλάξει. Και στα κρατημέλη μπορεί να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να βελτιώσουν τι επιδόσει των καταβολών. Τώρα για την ε, επίδοση και όπω η DG για την περιφερειακή πολιτική και εμεί ε, στην αρχή το 2014 ξεκινήσαμε σιγά σιγά αλλά τα πράγματα επιταχύνθηκαν για τον ρυθμό της ε, υλοποίησης και το Κοινωνικό Ταμείο και τον Ιούλιο του 17 φτάσαμε το 76% όσον αφορά το ποσοστό επιλογής και έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερη απορρόφηση, επιτάχυνση του ρυθμού απορρόφησης 26,2% τώρα. Δεν βοηθάει ο κανόνα του νη συν. Ε, και αυτό είναι το βασικό θέμα. Έτσι, παρακάμπτουν την πειθαργία που θα έπρεπε τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και κατέβηκε η απορρόφηση. Έπεσε. Δεν είναι όπως τη θέλαμε. Και όπως είπα και στην αρχή, να ολοκληρώσω λέγοντας κάποια ε, αριθμητικά στοιχεία που έχουμε όσον αφορά τα αποτελέσματα της δουλειάς μας με τα ταμεία. Είναι καλά τα μαντάτα, γιατί έχουμε πάνω από 26 εκατομμύρια Ευρωπαίων που έχουν βοηθηθεί από το Κοινωνικό Ταμείο και την πρωτοβουλία ε, απασχόλησης. Και έχουμε μεταξύ αυτών και 4 εκατομμύρια μικροφωνούς ανέργους. Όλα αυτά στην κρίση ε, που βοήθεια προς τον κόσμο και προς τα κρατη 2,6 εκατομμύρια που έχουν συμμετάσχει προγράμματα βρήκαν δουλειά, 3,6 εκατομμύρια απέξαν κάποιε δεξιότητε και 1,4 ε, εκατομμύρια ε, μπήκαν στην ε, παιδεία, στην κατάρτιση κατόπιν των δραστηριοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρωτοβουλία για απασχόληση των νέων απέδειξε ότι αξίζει και αυτό μα χαροποιεί. Γι' αυτό και η κυρία Φοντερ Λάιεν το έθεσε το ζήτημα ως προτεραιότητα θα τα ξανασυζητήσουμε με το που θα πάρουν το πράσινο φως αυτές οι προτάσεις ε, και σε πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό σας λέω ότι τώρα πρέπει να ολοκληρώσω και θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω σωστά τις ερωτήσεις σας. Και ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα διευθύνω εγώ τη συζήτηση στα ισπανικά. Ευχαριστούμε κύριε Κόρτε. Να δούμε τώρα τις ερωταπαντήσεις. Δεν έχουμε εδώ την εισηγήτρια. Ε, ο κ. Σοκόσκι θα κάνει τις ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Κόρτα για την εισήγηση και για τα όσα μας εξήγησε κάθε φορά. Είναι χαρά μας να ακούμε τις απόψεις σας Θέλω όμως ε, να σας κάνω πολλές ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις και μία εξ αυτών εξής. Ε, πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση απόδοσης αναφέρει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά το συνολικό ποσό που διακυβεύεται. Ε, μειώθηκε το γενικό ποσοστό σφαλμών, σφάλματος, ε, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως ε, στην βελτίωση της πολιτικής συνοχής. 1,1% ποσοστό σφάλματος, αυτό ήταν απλά μία πρόβλεψη και θέλω να ρωτήσω το Κοινοβούλιο Πώς ε, και εμπιστεύεται τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πώς είναι δυνατόν να υπολογίσει κανείς ε, τον κίνδυνο με βάση απλές ε, προβλέψεις. Και το δεύτερο ερώτημά μου είναι η εσωτερική υπηρεσία ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πώς μπορεί να εκδώσει μια θετική άποψη με βάση τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο MPR. Στη σελίδα 83 βλέπουμε, εκεί αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει έρθει σε διαβουλεύσεις, διαβουλεύσεις με το ελεγκτικό συνέδριο για να βελτιώσει το ποσοστό σφάλματος στο μέλλον. Ε, θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσα να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Ε, πολύ. ωραία. Η κυρία Πένκοβα. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Κορτέ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Εγώ θα επαναλάβω την ε, ερώτηση που έκανα και προηγουμένως. Υπάρχει το θέμα της απάτης. Μήπως ε, μπορείτε να μας προσφέρετε στοιχεία ε, για το θέμα της κοινή στρατηγικής για φέτος. και το δεύτερο ερώτημά μου είναι επίσης πολύ σύντομη. Ε, στην ετήσια έκθεση σας αναφέρεστε ε, στην ετήσια έκθεση για το κοινωνικό ταμείο. Εκεί περιλαμβάνονται στοιχεία του 2018 και αυτή η έκθεση ε, υπάρχει ήδη έκθεση εφαρμογής. Εστέλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο-τρεις γρήγορες ερωτήσεις. Πρώτον, για το κοινωνικό ταμείο. Στο παρελθόν κατηγορούσαμε τα κράτη-μέλη ότι δεν κάναν πολλές αξιολογήσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ενθαρρύνει η Κομισιό τα κράτη-μέλη να κάνουν συστηματικά αξιολόγηση του ταμείου αυτού, ώστε να εκπονούνται πολιτικές που να τεκμηριώνονται σε συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα. Δεύτερο, τι γίνεται με την εγγύηση για την νεολαία και άλλες προτάσεις για τη μείωση της νεανικής ανεργίας. Πρέπει και εδώ να έχουμε τα συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη πώς ε, παροτρύνεται για να παρακολουθούν την επάρκωση των τη συνέχεια τη εκθέσει, ποιότητα δεδομένων ε, για την εγγύηση για την νεολαία και για την απασχόληση των νέων. Και η βιωσιμότητα των επενδύσεων στα διευθυντικά ταμεία, πώς μετράτε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φουνκρά. Well, um, Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να επαναλάβω την ερώτηση που ήδη ετέθη για μένα. Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το εξή. Υπάρχει ένα προφανές γεγονός ότι ε, ορισμένα προγράμματα είναι περίπλοκα ε, και στην εφαρμογή και δεν μπορούμε να φτάσουμε στους πιο ευάλωτους. Γι' αυτό λοιπόν ε, όταν ακούω συγκεκριμένες απόψεις να εκφράζονται για το νέο σε δημοσιονομικό πλαίσιο και ότι θέλετε να βελτιώσετε τα κριτήρια για τα προσωπικά δεδομένα, ε, κυρίως ε, για τους ε, μακροχρόνια άνεργους και για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Από τη δική μας την εμπειρία θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να φτάσει κανείς σε αυτές τις ομάδες που ε, έχουν ειδικέ ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν είμαι καθόλου σίγουρη μήπως αυτό είναι πρόβλημα της Γερμανίας και των Γερμανών ή μήπως ε, το συμμερίζονται και άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να προειδοποιήσω σχετικά με τα κριτήρια και τα εμπόδια που μπορεί να υπάρξουν για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και ίσως ε, να έχετε κάποιες συγκεκριμένε απόψεις. Από τη μια προφανώς χρειαζόμαστε αντικειμενικά κριτήρια και πρέπει να αξιολογήσουμε τη διαδικασία. Από την άλλη, ε, κυρίως ε, για εκείνες τις ομάδες που έχουμε εμείς κατά νου, κάτι τέτοιο θα ήταν περισσότερο βάρος από το να είναι πρόσδεκτο. Σας ευχαριστώ Λούσα, για τις ερωτήσεις σας. Απαντήσεις παρακαλώ κύριε Κόρτε. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις ε, ερωτήσεις ε, και θα ήθελα να τις πάρω με τη σειρά. Ε, στην πρώτη ερώτηση, κύριε Τζερεχόφσκι, Κοιτάξτε, αυτά που ρωτήσετε είναι θέματα που μας απασχολούν και μένα προσωπικά πολύ. Ε, πράγματι, ε, θέσατε τον δάκτυλο σε πολύ σημαντικά θέματα. Το ποσοστό σφάλματος υπολογίζεται από το ελεγκτικό συνέδριο και από εμάς. Άρα, επ' αυτού έχετε δίκιο και σας συγχαίρω που το εντοπίσατε. Δεν το περίμενα, αλλά πολύ καλά κάνατε. Ε, αυτό είναι κάτι πολύ προβληματικό και πάει πίσω σε μία ε, διαφορετική μέθοδο που ακολουθεί ε, το ελεγκτικό συνέδριο, διαφορετική από αυτή που ακολουθούμε εμείς. διαφορετική λοιπόν μέθοδος και κάτι πρέπει να κάνουμε. Και το θέμα δεν είναι ότι θέλουμε να έρθουμε σε σύγκρουση με το ελεγκτικό συνέδριο ή εκείνη με εμά. Ε, το θέμα είναι πολύ πιο βαθύ και γι' αυτό θα ήθελα να ενθαρρύνω το Κοινοβούλιο να ε, θέσει το θέμα αυτό και στο ελεγκτικό συνέδριο. Εγώ είμαι ε, αρμόδιος για το ESF και για άλλα ταμεία και στην ετήσια έκθεσή μου πρέπει να αναφέρω τους κινδύνους για ένα συνολικό ημερολογιακό έτος. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Και αυτή η έκθεση που είδατε ε, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δουλεύω σε ημερολογιακή βάση, ε, θα πρέπει ε, να υπολογίσω τους κινδύνους για το δεύτερο εξάμεινο, αλλά δεν έχω στοιχεία. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Γι' αυτό με τους συναδέλφους μου κάνω μία πρόβλεψη που τη στηρίζω. Δεν έχω πρόβλημα να την υπερασπιστώ. Ε, την κάνω μαζί με τους συναδέλφους μου. Έχουμε αυτόν τον κανόνα του 10% που σημαίνει ότι για κάθε έτοιμα ε, κρατάμε ένα 10%, το βάζουμε κατά μέρος ε, και μόνο όταν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία ε, αποδεσμεύουμε αυτό το 10%. Άρα αυτό είναι ήδη μια άμυνα που έχω στα χέρια μου, δυνατότητα να αμυνθώ. Μετά, κάτι άλλο. Τα στοιχεία του παρελθόντος το ελεγκτικό συνέδριο έχει κάνει κατά το παρελθόν ε, μελέτες, ε, συζητάμε μαζί τους και τους λέμε ότι αυτό το θέμα δημιουργεί σύγχυση σε εσά και σε πάρα πολλούς άλλους. Φοβάμαι ότι δεν έχω λύσει επ' αυτού, αλλά θέλω να ελπίζω με την απάντησή μου σας εξήγησα ε, ποιο είναι το βασικό θέμα και πρέπει στο μέλλον να προσπαθήσουμε να έχουμε πιο αρμονικό υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος, κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο. Επίσης, είχατε ένα ερώτημα. Βασικά, όχι, νομίζω απάντησα στην ερώτησή σας. Αλλιώς μπορούμε να επανέλθουμε αργότερα. Η κυρία Πένκοβα σχετικά με τον αγώνα κατά τη, του, της απάτης και τη στρατηγική μας. Εγώ δεν νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει. Επεξεργαζόμαστε μαζί με τις άλλες γενικές διευθύνσεις ε, την κοινή μας ε, στρατηγική κατά της απάτης που συνεχίζεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ενέκρινε αυτή τη στρατηγική τον Απρίλιο του 2019 και νομίζω ότι πολύ σύντομα ε, θα μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε την κοινή στρατηγική για τα διαρθρωτικά ταμεία. Και πάλι η βασική ευθύνη, όποια στρατηγική και αν εφαρμόσουμε, ε, αφορά τα κράτη-μέλη. Αλλά δουλεύουμε ενεργά μαζί τους και καλούμε τα κράτη-μέλη να δουλέψουν σκληρότερα και κυρίως να ενισχύσουν τα αναλυτικά εργαλεία και για την ε, προδραστική ανάλυση του κινδύνου απάτης. Εδώ έχουμε το σύστημα αράκνε, αράχνη, που βασίζεται στις ε, διασυνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους ε, διάφορους ε, επιχειρηματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα αλγόριθμο που τα συγκεντρώνει όλα αυτά και έτσι μπορούμε και εμείς να κάνουμε μια πολύ χρήσιμη ανάλυση για το πού ακριβώς βρίσκονται κίνδυνοι απάτης ε, των, για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτό το σε πολλές περιπτώσεις μαζί με τα κράτη-μέλη. Ε, ένα στοιχείο της ε, στρατηγικής κατά της απάτης είναι να ε, χρησιμοποιεί αυτά τα αναλυτικά εργαλεία. Αλλά ο συνήθως όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε μαζί με τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα στην έκθεση εφαρμογής Νομίζω ότι σας ανέφερα ήδη κάποια στοιχεία για το τι κατά την άποψή μας έχει επιτευχθεί. Μέχρι το 16, 17, 18 πήγε πολύ καλά η εκτέλεση των προγραμμάτων. Και αν δούμε πιο συγκεκριμένα ε, για το ESF, τις προτεραιότητες, το 78% έχουν επιτύχει τους στόχους, το 20% δεν πέτυχε τους στόχους ε, και για δύο προγράμματα σε δύο κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν μπόρεσε να καταλήξει στο αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι γιατί τα στοιχεία που δόθηκαν δεν ήταν αξιόπιστα. Κύριε αν μου κάνετε μια ερώτηση για τη σημασία των αξιολογήσεων, Έχω συμφωνώ. Και στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ μου υπάρχει ομάδα που ασχολείται μόνο με αυτό, με τις αξιολογήσεις. Άρα μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως έχει μείζωνα σημασία για μένα το θέμα των αξιολογήσεων. Προσπαθούμε πάντοτε να παίρνουμε περισσότερες πληροφορίες, να βελτιώνουμε τα εργαλεία μας και συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη για να μπορούμε να αξιολογούμε τον πραγματικό αντίκτυπο των προγραμμάτων μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το ίδιο ισχύει για την πρωτοβουλία για τους νέους. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά βρέθηκαν αδυναμίες σε κάποια κρατημέλη, οι οποίες εντοπίζονται ακριβώς στην παρακολούθηση ε, των συμμετεχόντων. Δηλαδή, αν μπορούμε πραγματικά να αποδείξουμε ότι κάποιος που συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα, εν συνεχεία, είτε κρατάει τη θέση του, είτε συνεχίζει την εκπαίδευσή για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων. Πολύ καλή ερώτηση και αυτή ίσως σημαντικότερη για τους συναδέλφους ΓΔ Ρέτζιο, διότι εμείς κάνουμε επενδύσεις στις δομές, υποδομές, συγγνώμη. Εμείς μιλάμε για άτομα, για πρόσωπα. Παρακολουθούμε, λοιπόν, τα άτομα αυτά, τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν βρει μια δουλειά, μια θέση κάπου. Και προσπαθούμε επίσης να κάνουμε και μια αναφορά σε σχέση με τον αριθμό των ετών που έχουν κρατήσει αυτή τη θέση. Το θέμα είναι να βγουν από την ανεργία. Αυτό είναι ο βασικός σκοπός. Και τέλος ε, υπάρχει ένα ερώτημα ε, σχετικά με τη δυσκολία που υπάρχει το να έχουμε ε, αποτελεσματικότητα για τους πλέον ευάλωτους της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αυτό είναι αλήθεια. Η γενικότερη εικόνα ε, όσον αφορά ε, στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε γενικές γραμμές είναι καλή. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ενεργοί πολίτες είναι 241 εκατομμύρια. Αυτά, αυτός είναι ο υψηλότερος αριθμός από εποχής πρώτης καταγραφής των εργαζομένων. Ε, βεβαίως, προφανώς, αυτές οι θέσει έχουν φτιαχτεί όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τι επιχειρήσει. Πάντω η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Ε, και αν δείτε πόσοι άνθρωποι από ευάλωτε ομάδε βγήκαν από τη φτώχεια και βρήκαν δουλειά, ε, είναι εντυπωσιακό ο αριθμό. Παρ' όλα αυτά είναι εξίσου σαφές ότι αν πάει κανεί πέρα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πολύ καλός, ε, ε, βλέπει ότι υπάρχουν πολλοί θύλακες ε, προβλημάτων σε πολλά κράτη-μέλη. Το ποσοστό ανεργίας ε, των νέων στη δική μου χώρα, ας πούμε την Ολλανδία, είναι 3 ή 4%, κατ' ουσίαν δεν υπάρχει, αλλά σε άλλες χώρες, σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, εκεί τα ποσοστά είναι δεκαπλάσια. Άρα δηλαδή πράγματι το θέμα πρέπει να επανεξεταστεί και γι' αυτό νομίζω ότι το ε, μήνυμα που ξέπεμψε η υποψήφια πρόεδρος είναι πάρα πολύ καλό. Και άλλες ομάδες, η Ρωμά, η Βιβί, η συνάδελφός μου θα μιλήσει γι' αυτό. Ε, συνεργαζόμαστε με τους Ρωμά και με τους μετανάστες ε, για να μπορούν να εγκατασταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και αυτή είναι μια πολύ ευέλικτη ομάδα. Και αυτή είναι μια δουλειά ε, που ελπίζω θα μπορέσουμε να την προχωρήσουμε κατά την επόμενη θητεία μας και με τη δική σας υποστήριξη. Ευχαριστούμε τώρα Γενική Διευθύντρια για θέματα μετανάστευση ιστορικών υποθέσεων, κυρία Μίχου. Έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας για την παρουσίασή σα. Uh, Καλησπέρα σας και ευχαριστώ Πρόεδρε και κύριοι βουλευτέ και κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ και πρόκειται να έχουμε έναν διάλογο ανοιχτό για τις δραστηριότητε της Γενικής μας Διεύθυνσης το 18. Οπότε και πρόκειται για την πρώτη μου χρονιά ως Γενικής Διευθυντρίας και σας διαβεβαιώνω ότι δουλέψαμε σκληρά. Μια αποφασιστικότητα ούτως ώστε να μπορέσουμε με τις πολιτικές που ασκήσαμε να λύσουμε τα προβλήματα, να συντονίσουμε τις προσπάθειες σε όλα τα μέτωπα. Για να έχουμε καινούργια συστήματα πληροφορική, να είναι διαλειτουργικά, να έχουμε οικονομική, επικοινωνική βοήθεια για να μπορέσουμε να έχουμε υλοποίηση των μέτρων για ασφάλεια και μετανάστευση. Και να σας πω δύο λίγων ότι πετύχαμε την πολιτική μας στην μετανάστευση. Οπότε και συμφωνήσαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο. Όσον αφορά την ακτοφυλακή με ευξημένες αρμοδιότητες για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη. Είπαμε να θεωρηθεί σχετική οδηγία το νομικό πλαίσιο επίσης να αναβαθμιστεί το νομικό πλαίσιο για τις θεωρίες διαβατηρίων την ε, συνομοθέτηση επομένως αυτού του πλαισίου και τα σχετικά με το σύστημα VIS και η αυτή την πολιτική που υλοποιούμε σημασία έχει το να αποσπώνται συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το 2018 οι παράνομες αφήξεις εμειώθησαν. Κατέβηκαν στις 150.000 περίπου. Το οποίο ε, αγγίζει τα επίπεδα προ-κρίσεως. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα χειροβιαστό παράλληλα αυτά. Όμως, η κατάσταση είναι ευμετάβλητη και όπως θα πούμε αργότερα τους πιο πρόσφατους ε, μήνες, σε ένα-δύο διαδρόμους, έχουμε μία ελαφρά αύξηση. Αν των 25.000 έχουν μετεγκατασταθεί από τους πιο ευάλωτους μετανάστες και αυτό γίνεται με τα ταμεία της Γενικής μας Διεύθυνσης. Το 18 το Ταμείο Ένταξης Μετανάστευσης Ασύλου βοήθησε πάνω από 40.000 ούτως ώστε αυτοί να επαναπατριστούν σε σχέση με 16.000 το 17. Όμως, χρηματοδοτήσαμε τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αφήξεων, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, Μάλτα και Κύπρο. Αλλά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν πετύχαμε πάντοτε αυτό το οποίο θέλαμε. Γνωρίζετε ποιες είναι οι δυσκολίε όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου. Θα πρέπει να εξεύρουμε τρόπο ούτω ώστε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο και προσβλέπουμε στο Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει και επίσης η νέα πρόταση της Κομισιόν που έχει δεσμευθεί ε, τα είπε στις ενακτηρίες ομιλίες ε, ότι πρόκειται περί προτεραιότητας που έχει στον τομέα τη ασφάλειας. Η Γενική μα Διεύθυνση κατέβασε κάποιε νομοθετικέ προτάσεις, ούτω ώστε να καταπονημηθεί η τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα και στόχος ε, είναι να θωρακιστεί το πλαίσιο για τη θέση σε εμπορία των εκρηκτικών και διάφορες ποινικέ διαδικασίες και επίσης ε, για πάτες και για πλαστογραφία. Όλα αυτά πέρασαν το 19, αλλά ακόμη εκκρεμεί μια πρόταση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Η πρόταση που αφορά την διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο ίντερνετ. Και ελπίζουμε πάντως ότι οι συνωμοθέτε αυτό θα τον κρίνουν, θα τον κρίνουν σύντομα για τον προπολογισμό τώρα. Συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι πολιτικές μας είχαν πρικοδότηση 2,6 πιστώσεις ε, υποχρεώσεων και αυτό είναι το 2% του κοινωτικού προϋπολογισμού. Πάρα πολύ καλά ποσοστά εφαρμογής, υλοποίηση και απορρόφηση πάνω από 92% όσον αφορά τις πληρωμές και τις υποχρεώσεις και να ληφθεί η υπόψη η επίπτωση των ε, εισόδων, κάτι το οποίο αφορά τα δικά μας ιδιαίτερως ε, κονδύλια και καταφέραμε κατά 30% να μειώσουμε τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα προς, ε, προς, προς ανάλωση, παράλ, και ε, όλα αυτά παρακολουθήθηκαν στενά. Το ποσοστό απορρόφησης των κρατών για άσυλο, ένταξη, μετανάστευση και σε σχέση με την εσωτερική, εσωτερική ασφάλεια, του σχετικού ταμείου έχει ποσοστά ανωδικά Μικρό το ποστό κινδύνο, 17,7 εκατομμύρια και το σφάλμα είναι κάτω από το 2%. Οπότε το αποτέλεσμα αυτό είναι ακόμα πιο θετικό και ενθαρρυντικό σε σχέση με το συνολικό κόστος των ελέγχων μας που το 18 ήταν κάτω του αντίστοιχου ποσού του 17 παρά το ότι είχαμε περισσότερες πληρωμές το 18 ή στην έκθεσή μου υποβάλλω έξι επιφυλάξεις, δύο εξ αυτών. Μία, μία, μία εξ αυτών διορθώνει η μιλήτρια είναι νέα και αφορά την φυλακή εκτοφυλακή, τη νέα υπηρεσία. Για την υπηρεσία ασύλου παραμένει η επιφύλαξη και οι υπόλοιπε, οι υπόλοιπες 6 δηλαδή από τις επιφυλάξεις επίσης διατυπώθηκαν το 18 και αφορούν παλαιότερα κονδύλια για το αμύθ και το σόλτ. Οπότε ε, δύο έχουμε άρη για το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλη μία για το άμυθ και την Ελλάδα. Με αυτές τις επιφυλάξεις ε, φαίνεται ότι έχουμε δυναμική ενεργητική στάση και ότι οι διορθώσεις βοηθούν ούτως ώστε να υπάρχει ένα πνεύμα πρόληψης διότι έτσι οι δικαιούχοι και τα κράτη-μέλη ξέρουν ότι θα υπάρξει ανάκτηση των κονδυλίων όποτε χρειαστεί. Και εν κατακλείδη να σας πω τα εξή κυρίε και κύριοι και αξιότιμοι βουλευτέ. Η Γενική Διεύθυνση Ιστορικής Πολιτικής λειτουργεί με έναν ε, τρόπο δυναμικό σε ένα περιβάλλον πολιτικής το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς. Χρειάζεται συνεχώς προγραμματισμό για το μέλλον, αλλά επίσης ασχολούμαστε και με την ε, αξιοποίηση των κονδυλίων και έχουμε πάρα πολλές καταστάσεις κατεπήγοντες, οπότε πολλές φορές πρέπει να συμβάλλουμε στα εθνικά προγράμματα με επιπλέον χρηματικούς ε, πόρους και πόρους γενικά στο εσωτερικό, δε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, εύρυθμα λειτουργούμε, τόσο να υπάρχει συντονισμό για την χρήση των κονδυλίων σε εσωτερικό και εξωτερικό. Δεν ήταν πάντοτε εύκολα τα πράγματα και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έτσι ισχύει και πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ακόμα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά είμαι αποφασισμένη να συνεχίσω στην ίδια ρότα και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ούτως ώστε να μπορέσουμε μαζί να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Και σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ε, εμείς ευχαριστούμε κυρία Μίχου και τώρα έχουμε τον γύρο των ερωταπαντήσεων. Εσείς και σε είναι λίγο μπερδεμένο το όνομά σας. Δύσκολο να το βρω. Μια χαρά το είπατε το όνομά μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Μίχου για την παρουσίαση. Γνωρίζουμε ότι πολλά πράγματα ε, εξελίσσονται, πρόοδος υπάρχει, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική απόδοση. Ε, μη μας θυμώσετε πάντως ε, αν έχουμε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις για τη δική σας τη Γενική Διεύθυνση, διότι πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε πώς είναι δυνατά κάποια πράγματα, όπως το ζήτημα με το ΕΑΣΟ, παραδείγματος χάρη. Και έχουμε μια πολύ σημαντική ερώτηση για το πώς βλέπετε την ευθύνη της ΧΟΜ και τη δική σας ευθύνη στο θέμα της ΕΑΣΟ, γιατί σήμερα ψηφίζαμε για την απαλλαγή ε, της υπηρεσίας για το 2017 και με εξέπληξαν ε, τα αποτελέσματα της Όλαφ. Ε, επισκέφθηκα το καλοκαίρι την Άσο στο, ε, στις μου διακοπές και πραγματικά στη Μάλτα είδα πράγματα και θάματα να έχουν συμβεί. Πώς έγινε αυτό με μια τόσο μικρή υπηρεσία, είναι όνειδος είναι όνειδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ ε, δεν μπορούσα να φανταστώ στη ζωή μου ότι θα μπορούσε τόσο, ε, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κάνει κάποιος τόσα πολλά ε, πράγματα, σημεία και τέρατα, τόσα ασφάλματα, τόσα λάθη. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση, γιατί δεν έχει κάποιους βασικούς δείκτες επιδόσεων η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ό,τι αφορά την απόδοση του συστήματος ε, μεταγκαταστάσεων γιατί η γάμα Delta Home δεν έχει ε, βασικό δείκτη και performance indicator για την κατάσταση των πλέον ευάλωτων μεταναστών ιδίω παιδιών. Και μια πολύ σημαντική ερώτηση έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό. Eurojust και Europol αντιμετωπίζουν όλο και αυξανόμενο αριθμό υποθέσεων που μελετούν, ε, τις οποίες ασχολούνται. Θέλουμε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Eurojust, Europol, με όλα και άλλους φορείς. Όμως, το προσωπικό τους είναι λίγο και οι πόροι τους είναι λίγοι. Επίσης, εσείς ως γάμα τι κάνετε, πώς αντιμετωπίζετε την κατάσταση αυτή και ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον. Και μια άλλη ερώτηση. Τι προβλήματα εντοπίσατε σε Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο και στη Φιλανδία και στην Ελλάδα για το άμυφα και πριν για το Solid ε, και στις δύο προηγούμενες χώρες δηλαδή. Γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος ε, να διορθωθούν τα προβλήματα τα οποία από το 2013 έχουν διαπιστωθεί στη Γερμανία. Και σε ένα τελευταίο ερώτημα. Ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος των συνδέσμων, των liaison officers ε, για τη μετανάστευση και τι αξία πραγματική έχουν στην προσπάθεια που κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πένκοβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Θέλω να σα ευχαριστήσω κυρία Μίχου για την πολύ αναλυτική παρουσίαση. Έχω ένα πολύ σύντομο ερώτημα. Υπήρξε στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου 17 ε, μια σύσταση και η ΓΔΧ σε συνέχεια της σύστασης λέει ότι προετοιμάζει ένα guidance note, ε, οδηγία λοιπόν προς τα ε, κράτη-μέλη ό,τι αφορά το ΦΠΑ ε, που δηλώνουν οι δημόσιοι φορείς. Θα ήθελα να μας κάνετε μία ενημέρωση. Πού βρίσκονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες για αυτό το σημείο. Με ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σαστέλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Αρχικά, σε ό,τι αφορά τις επιφυλάξεις ε, για εμβληματικά προγράμματα της ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ όπως είναι το ΆΜΙΦ, ε, το Internal Security Fund, ε, όπου από το 14 έως 20 τον προϋπολογισμό ε, γίνεται λόγος για σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση και στο σύστημα ελέγχου. Θα ήθελα να μου πείτε τι μέτρα προβλέπετε για να ενισχύσετε τους ελέγχους σε σχέση με τα κράτη-μέλη Και θα ήθελα ε, μια σύντομη ανάλυση, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, Τι γίνεται με τη διευκόλυνση ε, για τη διαχείριση των ε, προσφύγων στην Τουρκία με ΜΚΟ κυρίως δηλαδή και πώς γίνεται η αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων τα οποία είναι διαθέσιμα και κάτι παραπάνω αν μπορείτε να μας πείτε για τη διαχείριση και τη λειτουργία των hot spot. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Επίσης, με ποιο τρόπο η δική σας Γενική Διεύθυνση συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες για τη βελτίωση της πολιτικής επικοινωνίας της Ένωσης σε ό,τι αφορά τα βασικά επιτεύγματα της πολιτικής της Ένωσης σε θέματα μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Φουκράου δεν τη βλέπω, δεν ξέρω αν θέλει ο κύριος Πέσκα να πάρει τη θέση της, να κάνει κάποιες ερωτήσεις, όχι. Οκ, okay. περνάμε λοιπόν στις απαντήσεις από την κυρία Μίχου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. to be angry for... Φυσικά και δεν θα σας θυμώσω για τις ερωτήσεις που μου κάνετε, διότι γνωρίζω ότι όσο και εγώ έτσι και εσείς ενδιαφέρεστε να βρεθούν λύσεις σε αυτόν τον τομέα πολιτικής που έχω την τύχη να καθοδηγώ. Ε, να είμαι υπεύθυνη αυτής της Γενικής Διεύθυνσης. Ε, ξεκινάω την ΕΑΖΟ. Γνωρίζω ότι σήμερα το πρωί αποφασίσατε να μην χορηγήσετε απαλλαγή για το 2017 και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας. Τα λέω έξω από τα δόντια. Ως γάμα Δέλτα Home έχω επιφύλαξη ε, για το 2017 για την ΕΑΖΟ ο νέος διευθύντης, η νέα διευθύντρια συγκεκριμένα ήρθε εδώ στο Κοινοβούλιο και εξέφρασε ε, ε, τις απόψεις της και είπε τι θα κάνει, αλλά για το 17 πρέπει να διαλευκανθούν τα πάντα. Και μετά θα άρω εγώ τη δική μου επιφύλαξη και εσείς θα μπορέσετε ενδεχομένως να άρετε τις δικές σας επιφυλάξει. Επομένως, τι μάθαμε. Εγώ εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως καταλαβαίνετε. Είμαι 16-17 μήνες στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Home και έφτασα ακριβώς στη στιγμή που είχα εργαστεί με την ΑΖΟ. Δεν θα πω τίποτα για τον εκτελεστικό διευθυντή. Μιλάω για το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ της ΑΖΟ και την Όλαφ. Είχα εργαστεί μαζί τους ώστε το συντομότερο δυνατό να μπορέσουμε να έχουμε την επόμενη μέρα για την υπηρεσία αυτή που είναι μια πάρα πολύ ε, νευραλγική υπηρεσία για τον τομέα στον οποίο εργαζόμαστε. Και μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο καταφέραμε ε, να ληφθούν διάφορα μέτρα που οδήγησαν στην απομάκρυνση του προηγούμενου διευθυντή ο εκτελεστικός διευθυντή. Ο εκτελεστικό διευθυντή, ο προσωρινό, ε, όρισε 250 ενέργειε. Μόνο το 10% ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί από αυτέ τι νέε δράσει ενέργεια. Και τώρα έχουμε την εκτελεστική διευθύντρια που δεσμεύτηκε που θα γίνει η εσωτερική έλεγχη ότι θα συνεργάζονται ο Γενικός Διευθυντής με τον εκτελεστικό διευθυντή και θα υπάρξουν σχέσεις καλές που θα μας εξασφαλίσουν πως αυτά τα οποία συνέβησαν δεν θα ξανασυμβούν. Από πλευράς μου. Ως Γενική Διευθύντρια. Έχω αλλάξει τα μέλη που συμμετέχουν στο ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ. Από τα μέλη της προηγούμενης χρονιάς η Γενική Διευθύντρια και αναπληρωτή συμμετέχουν στα ΔΕΛΤΑ Σίγμα. Have created in the Θέλω να σας πω ότι έχουμε αναδιαμορφώσει τη Γενική Διεύθυνση Home και εκεί υπάρχουν ομάδες οι οποίες δουλεύουν πολύ συγκεκριμένα για να παρακολουθούν τους φορείς και δεν μιλάω μόνο για την Αζό, μιλάω για, όλες, για όλους τους οργανισμούς. Όλη λοιπόν αυτή η δουλειά γίνεται έτσι ώστε ε, πρώτα απ' όλα να ξέρουμε τι συμβαίνει στις διάφορες, στις οργανισμούς, αλλά επίσης και για να υπάρχει στην Επιτροπή η γνώση που είναι απαραίτητη έτσι ώστε να μην ε, προκύπτει επικάλυψη εργασιών. Ε, να μην κάνουν όλοι οι οργανισμοί τα ίδια. Έτσι λοιπόν, ε, αν με ρωτάτε το τι σημαίνει τώρα στην ΕΑΖΟ, έχουμε εσωτερικά πρότυπα ελέγχου, Έχουμε ελέγχους και έρευνες, check and balance κατ' ουσίαν. Ε, έχουμε βελτιώσει τη συνεργασία ανάμεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Εκτελεστικό Διευθυντή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Γι' αυτό πιστεύω ότι εφαρμόζουμε σωστά τους διαγωνισμούς και τις ε, προσλήψεις και είμαι σίγουρη ότι ακολουθούμε, είμαστε καταδικασμένοι να ακολουθήσουμε τη σωστή κατεύθυνση. Ε, τώρα, όσον αφορά τα βασικά στοιχεία για την εγκατάσταση των μεταναστών. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα μέχρι το 2020 δεν έχει λάβει υπόψη του τις ε, ειδικέ ε, ανάγκες που έχουμε τώρα μετά το 2015 και το 2016 και γι' αυτό το λόγο κάναμε το εξής. Έχουμε πολλές εκθέσεις ε, που αφορούν στην επαναγκατάσταση, στην επαναπροώθηση, ε, ανθρώπους που είναι ευάλωτοι, ε, μετανάστες που είναι επιλέξιμοι και άλλοι όχι πόσοι έχουν ενσωματωθεί. Η απάντησή μου λοιπόν είναι ότι έχουμε πολύ αυστηρό έλεγχο της κατάστασης, έχουμε επανειλημμένα ε, αναφερθεί στην πρόοδο και την έλλειψη συγκεκριμένων δικτών ε, απόδοσης την έχουμε εντάξει στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που διαπραγματευόμεθα με εσά και το Συμβούλιο. Η Europol, η Eurojust, τα προγράμματά μας για το μέλλον. Η Europol είναι κάτω από τη δική μου τη Γενική Διεύθυνση. Η Eurojust είναι στη Γενική Διεύθυνση Justice, δικαιοσύνη. Εγώ έχω έξι οργανισμούς, η Europol είναι ένας από αυτούς και η Europol μετά το 2015 τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι άλλαξε τελείως ο ρόλος της ε, Europol. Η εντολή πλέον της ε, Europol είναι ε, η αξιολόγηση του 2021. Εν τω μεταξύ έχουμε προσπαθήσει ως Επιτροπή να στηρίζουμε πάντα τη Europol διότι τους έχουμε δώσει πολλά νέα καθήκοντα λόγω των ε, αναγκών που έχουν προκύψει από το 2015 μέχρι σήμερα. Και η Europol ε, προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, αν υπάρχει κάποιος που στηρίζει τη Europol για να ε, καλύπτει τις αρμοδιότητές της, τότε αυτή είναι η δική μας, η Γενική Διεύθυνση και βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά ε, κοιτάξτε κι εγώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι αν δεν έχω τη νομική κατοχήρωση, δεν μπορώ τώρα να αλλάξω την εντολή της Europol. Ε, διότι υπάρχουν κάποιες ε, ελλείψεις ε, από το 2015 μέχρι σήμερα. Όμως το έχουμε μάθει το μάθημά μας και ελπίζω με τη δική σας την υποστήριξη θα κατορθώσουμε στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να έχουμε μια Europol η οποία θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Παραδείγματο χάρη τους ε, ζητάμε να είναι για μας ε, ένας φορές που θα μας παρέχει πληροφορίες, να εργάζονται για την διαλειτουργικότητα, για τις επαφές ε, των ε, τρομοκρατών ηλεκτρονικά. υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και χρειάζονται γι' αυτό να δοθούν και κονδύλια. Γιατί τόσο πολύ διήρκησε μέχρι να έρθουν επιφυλάξει. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ όλα αυτά να γίνουν μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε εμά και τα κράτη-μέλη. Και πέρυσι έκανα την ίδια ερώτηση και μου έδειξαν πόσες ανταλλαγές έχουμε με τα κράτη-μέλη για να κατανοήσουν τι είναι απαραίτητο και σε τελική ανάλυση ε, όταν έρωμη επιφύλαξη, αυτό το κάνω, είτε διότι το σύστημα του κράτους μέλους δεν λειτουργήσε καλά, είτε διότι πήραν χρήματα, είτε διότι εντοπίστηκαν κάποιες άλλες ελλείψεις σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι λοιπόν εύκολο να ε, κάνω πολύ γρήγορα όλες αυτές τις ε, διορθώσεις. Όπως είπα στην εισαγωγή μου, ε, συνεργαζόμαστε στενά με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξη ε, για να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις της μετανάστευσης και στο ιστορικό και στο εξωτερικό. Και βεβαίως έχουμε και τις αντιπροσωπείες μας. Και οι αντιπροσωπείες μας δίνουν και μέσα από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης μας δίνουν τις πληροφορίες ε, που χρειαζόμαστε για τις ε, τρίτες χώρες. Όμως αντιμετωπίσαμε πέρυσι ένα πρόβλημα. Παραδείγματο χάρη, εμείς θέλαμε για ε, τις οικειοθελείς επιστροφές να έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για υπηκόους τρίτων χωρών. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό ήταν δύσκολο να γίνουν οι σωστές επαφές με τις τρίτες χώρες. Και εμείς ε, χωρίς ε, τους ανθρώπους που τώρα όμως τους έχουμε και βλέπω εδώ ότι έχουμε 11 στην Ιορδανία, Μαρόκο, ε, Σερβία, Σουδάν, την Ισία, Νίγηρα και αλλού, στο Μπαγκλαντές, στην Αίγυπτο, στην Τουρκία Μπορέσαμε λοιπόν να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας ε, για να μπορέσουμε να αποκτούμε ε, καλύτερες διαδικασίες, γρηγορότερες, να αποκτάμε πληροφορίες ε, για τις τάσεις, για την έγκαιρη προειδοποίηση. Έχουμε αναφορές. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ε, ε, εφαρμογή προγραμμάτων ε, με τρίτες χώρες για την πολιτική επαναπρόθεση. και προσπαθούμε και να βελτιώσουμε <coughs> την κατάσταση. Έχουμε το δίκτυο που αφορά όσους εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και για τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά στο ερώτημα σχετικά με το ΦΠΑ, έχουμε ζητήσει από τα κράτη-μέλη να ε, συμπληρώσουν ε, ένα ερωτηματολόγιο. Αυτό θα γίνει μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Με βάση αυτό θα αξιολογήσουμε τις ανάγκες. Ε, μετά το Σεπτέμβριο θα μπορώ να σας πω πώς θα προχωρήσουμε. όσον αφορά στις τάσεις για την Τουρκία και ποια είναι η κατάσταση με εκείνους που έχουν να ε, διαπραγματευτούν με την Τουρκία της Μίκιο. Η κατάσταση δεν είναι τόσο εύκολη, αλλά στον τομέα της μετανάστευσης έχουμε αποτελέσματα. Γνωρίζουμε ότι ισχύει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και οι αφήξεις ε, μέχρι και πριν από 15 ημέρες στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη δεν ήταν ε, ιδιαίτερα μεγάλες. Μείωση κατά περίπου 90%. Σήμερα όμως διαπιστώσαμε τουλάχιστον τις τελευταίες ε, εβδομάδες ότι έφτασαν περίπου 7 με 8.000 άνθρωποι. Ε, τώρα, στην Τουρκία έχουμε 4 εκατομμύρια και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τα κονδύλια που διαθέτουμε, κυρίως ε, στους εταίρους μας τα διαθέτουμε, αυτά ε, αποδίδουν. Δεν έχω να ακούσει τώρα να υπάρχει πρόβλημα που να αφορά στις σχέσεις ε, της Τουρκίας ε, με τους εταίρους μας. Αυτό υπήρχε πέρυσι, αλλά τώρα η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται μάλλον για το 24.000 Σύριοι οι οποίοι επαναγκαταστάθηκαν ή επαναπροωθήθηκαν. Και ενώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, είναι τα μάτια μας ανοιχτά, να βλέπουμε τι συμβαίνει στην Τουρκία, παράλληλα οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα σε όλες τις ε, πτυχές ε, της συμφωνίας. Τώρα, η διαχείριση των καταβλισμών, των hotspot. Συγγνώμη, μπορείτε να τελειώσετε. Ξέρω ότι μακρηγορώ και είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε μετά να συζητήσουμε. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση στους καταβλισμούς στην Ελλάδα, δεν είναι καλή και ε, διαθέτουμε κάποια κοντήλια Η κατάσταση βελτιώνεται. Η κατάσταση βελτιώνεται κάθε ημέρα που περνάει. Σύντομα θα έχουμε χειμώνα. Η κατάσταση σχετικά με τους ασυνόδευτους ε, ανήλικους ε, υπάρχει μια στρατηγική. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αν φτάνουν σε ένα καταβλισμό 7.000 άνθρωποι την ημέρα, πρέπει να έχουμε τις δυνατότητες, ε, τις οικονομικές και άλλες, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις ελληνικές αρχές να αντιμετωπίσουν ε, αυτό το πρόβλημα. Και ζητάμε, έχουμε καταρτήσει προγράμματα δράσης για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα σε καθημερινή βάση. Τώρα πώς επικοινωνούμε αγαπητοί ευρωβουλευτές και θα τελειώσω με αυτό. Έχουμε κάνει πάρα πολλά. Και ακούγοντας όμως τα μέσα ενημέρωσης, αν υπάρχει κάτι αρνητικό, αυτό λένε, αυτό προτείνουν και προβάλλουν. Τα καλά δεν τα λένε. Ο δικός μου λοιπόν ο ρόλος ε, ως υπαλλήλου, ανώτατο υπαλλήλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με άλλους συναδέλφους, είναι να διασφαλίσω ότι τα κονδύλια που διαθέτουμε ε, δαπανώνται σωστά, ότι η πολιτική που εφαρμόζουμε ε, αποδίδει και σε τελική ανάλυση αντιμετωπίζουμε τις ε, ενστάσεις και στην μετανάστευση και στην ασφάλεια. Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό υπάρχουν πλέον λιγότερα προβλήματα για τους πολίτες. Είναι όμως δύσκολα τα πράγματα, μπορούμε να βελτιωθούμε, κάνουμε πάρα πολλά και το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι χρειάζομαι την υποστήριξή σας για να περάσουν σωστά μηνύματα. Και ελπίζω ε, πλέον με τη νέα Επιτροπή θα μπορέσουμε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και επικοινωνίες. Ευχαριστώ. Οι διερμηνοί σας ενημερώνουν ότι η διερμηνία δυστυχώς εδώ πρέπει να σταματήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Señor Duens, tiene cinco minutos para la primera exposición. Vamos a intentar ir lo más rápido posible porque el servicio de interpretación también tiene que, que irse. Gracias.